Uh, Συνάδελφοι, έχουμε μια επίκαιρη συζήτηση τώρα, την κατάσταση στην Ιγυρία και θα ήθελα να καλωσορίσω τον καρδινάλιο Τζον Ολουρφέμιο Ναγέκαν, που είναι οραμακαθολικός καρδινάλιος και αρχιεπίσκοπος της Αμπούζα. Σεβασμιότατε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ εκπρόσωπος της ε, Ρωμαϊκής Εκκλησίας, μία από τις πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, η οποία συντίθεται από πολλές εθνότητες ε, και θρησκείες και χαρακτηρίζεται και από το δέλτα του Νίγηρα όπου παρουσιάζονται πολλά προβλήματα ε, από ακραίες Ισλαμιστικές οργανώσεις στο Βορρά. Το Σύνταγμα της χώρας εγγυάται την ε, ε, ελευθερία πίστης, ανεξιθρησκεία δηλαδή, και ενώ στο Βόρα έχουν εισαγάγει τον ε, ε, Ισλαμικό νόμο της ε, Σαρία. Υπάρχουν, γίνονται συγκρούσεις και υπάρχουν και πειρές της Αλκαΐντα μέσω του Ισλαμικού Μαγκρέμπ. Η Νιγηρία έχει επικριθεί για μια πολύ σκληρή αντιμετώπιση και έχει επικριθεί ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα εφαρμόζοντας ε, αποφάσεις εκτός ε, του διεθνούς δικαίου και ε, επίσης το πολιτικό κλίμα πριν από τις εκλογές του 2015 χαρακτηρίζεται από μεγάλες εντάσεις και αυτήν την έντονη διαίρεση μεταξύ Βορρά και Νότου. Σε θα μας δώσει η ανταλλαγή αυτή των απόψεων και η σημερινή συζήτηση την ευκαιρία να ενημερωθούμε καλύτερα για το τι συμβαίνει στη χώρα και το τι προσδοκίες έχετε για την υγεία σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας εδώ και αναμένουμε ε, την ε, εισήγησή σας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Καταρχάς, ευχαριστώ τους διοργανωτές της ε, σημερινής συζήτησης και που μου έδωσε την ευκαιρία να αποτανθώ σε αυτό το εξέχον σώμα. Ε, ε, και ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δώσατε. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω αυτή την επιτροπή που βρήκε το χρόνο να με προσκαλέσει και να με ακούσει. Γνωρίζω ότι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σώμα και εκπρόσωπος εθνών έχει, έχει πολλές πηγές από τις οποίες ενημερώνεται για τη χώρα μου την Νιγηρία και πρέπει να πω ότι η σύντομη περίληψη που κάνατε κύριε Πρόεδρε ε, δείχνει ότι είσαστε πολύ καλά πληροφορημένοι για τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μου. Γνωρίζω ότι τα κράτη σας έχουν πρεσβεία στην Αμπούτζα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ε, την εκπροσώπησή της. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω ε, την πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έτσι γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο. Επίσης γνωρίζουμε την ε, κάλυψη των προβλημάτων της Νιγηρίας από τα μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς πρέπει να πω και αυτό είναι λυπηρό ότι τα νέα που προέρχονται από τη χώρα μου είναι πάντοτε αρνητικά στον τύπο, στα μέσα ενημέρωσης και δεν λένε τίποτα για τις προσπάθειες που γίνονται να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Υπό το φως λοιπόν αυτών των γεγονότων θα ήθελα μέσα στα 7 με 10 λεπτά που έχω χρόνο ομιλίας να παρουσιάσω την άποψή μου ε, από την οπτική γωνία ενός θρησκευτικού ηγέτη και δι ε, Ρώμα καθολικού καρδιναλίου που έχει ζήσει στην Ιγυρία πολλά χρόνια αποτελώ λοιπόν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας, της μάχης που δίνουμε εκεί με την συνεχώς ε, εναλλασσόμενη κατάσταση συνθήκων ε, και πραγματικότητος. Ε, τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν και εξελίσσονται ε, και βεβαίως ε, είναι γνωστό ότι η Νιγηρία έχει μια μεγάλη ποικιλία ε, θρησκειών αλλά βασικά στο εθνικό επίπεδο είμαστε μισή χριστιανοί, μισή μουσουλμάνοι. 60 από τα... However, από τα 260 εκατομμύρια περίπου η μισή είναι χριστιανοί, η μισή είναι μουσουλμάνοι. Some parts of the... Και το αποτέλεσμα είναι, επειδή η γεωγραφική κατανομή δεν είναι ακριβώς ισομερής, ε, υπάρχουν περιοχές όπου βασικά επικρατεί χτενική θρησκεία στον πληθυσμό και σε άλλες περιοχές επικρατούν οι μουσουλμάνοι, η μουσουλμανική θρησκεία. Αλλά καμία περιοχή δεν είναι αμυγός ή το ένα ή το άλλο. Πάντοτε υπάρχουν και οι δύο θρησκείες. Άρα λοιπόν ε, αυτό δείχνει ότι πρέπει να συνεπάρξουμε και πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί. Και πιστεύω ότι αυτό ισχύει σήμερα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της Ισλαμικής τρομοκρατίας που πιστεύω σας απασχολεί ιδιαίτερα και απασχολεί και μένα. Η χώρα μας είναι περίπλοκη και ε, μου θυμίζει το μύθο των 10 τυφλών ανθρώπων που πήγαν να δουν τον ελέφαντα όπου ο καθένας άγγιξε ένα μέρος του σώματος του ελέφαντα και έτσι διαμόρφωσε μια διαφορετική εικόνα αν θέλετε επειδή ήταν τυφλή ε, της εικόνας του ελέφαντα. Έτσι περίπου αυτό ισχύει και για την Ιγυρία. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές απόψεις, τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις που τώρα έχουμε καταλήξει ότι δύο μεγάλες προκλήσεις είναι η διαφθορά και η ανασφάλεια. Δεν είναι καινούργια προβλήματα αυτά, αλλά είναι τα πιο εξέχοντα. Είναι τα πιο σημαντικά σήμερα. Και τα δύο αυτά προβλήματα είναι πρόκληση μεγάλη για την διακυβέρνηση της χώρας. Μία διακυβέρνηση η οποία ακόμα είναι αστασής και δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την αξία της. Δεν θα πω πολλά για τη διαφθορά, είναι πασίγνωστα όλα αυτά, ε, υπάρχουν ε, αξιωματούχοι επίσημοι, κυβερνητικοί δηλαδή, που είναι διεφθαρμένοι και πολλές φορές τη διαφθορά αυτή μένει ατιμόρυτη. Ε, ε ίσως πολλές φορές είναι και νόμιμη μάλιστα. η κυβέρνηση αναφέρεται σε αυτό το, το κακό, έχει δημιουργήσει μια ειδική ομάδα κατά πολέμηση της διαφθοράς, αλλά περιμένουμε ακόμα να δούμε πώς θα ξεριζώσει αυτό το φαινόμενο. Διότι εμείς ως θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να δούμε πώς θα ε, ξεφύγουμε από, αυτήν την, από την, ε, από αυτό το πρόβλημα, από τα δεινά, διότι έχουν και πνευματικές επιπτώσεις. Δεν είναι μόνο οικονομικές και πολιτικές, αλλά και πνευματικές επιπτώσεις στην, ε, στο ηθικό. Τώρα, το άλλο μεγάλο πρόβλημα. Όπως ε, ξέρετε υπάρχουν διαφορές μέσα στη χώρα μου, διαμάχες του παρελθόντος, αυτό βεβαίως ισχύει και στις χώρες της Ευρώπης διαμέσου των αιώνων. Είχαμε λοιπόν ε, διαμάχες ε, μεταξύ μειονοτήτων στη χώρα μας ε, όπου μία φυλή πολεμούσε την άλλη πριν από την απεικιοκρατία μάλιστα και πολλές από αυτές τις έχθρες υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Επίσης έχουμε ποινικά αδικήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται και επίσης θρησκευτικέ σειράξεις όπου μέλη μιας ενός δόγματος εμπλέκονται σε αιματηρές σειράξεις. Πολλές από αυτές τις σειράξεις και στο παρελθόν δεν ήταν καθαρά θρησκευτικά, θρησκευτικές, αλλά προέκυψαν από χειραγώγηση ε, του πληθυσμού, από, διάφορες, ε, ε, από διάφορους θρησκευτικούς αρχηγούς που είχαν τους δικούς τους ιδιωτελείς σκοπούς και ήθελαν να φέρουν σε αντίθεση και σύραξη τη μία φυλή εναντίον της άλλης, τη μία ομάδα εναντίον της άλλης. Υπάρχουν λοιπόν και πιο βαθιές ε, ρίζες αντιθέσεων και σειράξεων οι οποίες καλύπτονται με την επίφαση της θρησκευτικότητα. Δυστυχώς η αυτές οι θρησκευτικές διαφορές είναι πάρα πολύ ισχυρές. Μπορούν να επιφέρουν πολλά καλά, πολλά θετικά στοιχεία αλλά και μεγάλα δεινά όταν χρησιμοποιούνται κακώς οι προσπάθειες των θρησκευτικών αρχηγών δείχνουν ότι προσπαθούμε να εξασκήσουμε την πίστη μας, τη θρησκεία μας με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουμε μέρος της λύσης και όχι μέρος των προβλημάτων, αιτία προβλημάτων ε, και της ε, αιτία της ρίζας του κακού. Γι' αυτό ακριβώς ε, θέλω να μιλήσω για την ειδική περίπτωση της δραστηριότητα των Ισλαμικών τρομοκρατικών ομάδων, ιδίω στην βόρειο-ανατολική περιοχή της Νιγηρίας, αλλά όχι μόνο εκεί, και σε άλλες ε, περιοχές της χώρας, ε, σε ορισμένες χρονικές περιόδους. Αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο Ομολογώ ότι μας, μας βρήκε απροετοίμαστους και εκπλαγήκαμε, εκπλαγήκαμε. Ε, δεν περιμέναμε τέτοιου είδους ε, δρομοκρατικές ενέργειες, ε, βόμβες αυτοκτονίες βομβιστές αυτοκτονίας, ενδοφιλετικές ε, δολοφονίες, τρομοκρατικές απειλές ε, και ο στόχος αυτών των ακραίων ομάδων, το έχουν δείξει δηλαδή, είναι να γίνει όλη η Νιγηρία μουσουλμανική ε, και ε, ένας από τους στόχους τους βεβαίως είναι οι χριστιανικοί πληθυσμοί και τα, οι, οι επιχειρήσεις, η ζωή τέλο πάντων των χριστιανών και τα συμφέροντά τους σε δυσανάλογο ποσοστό. Έχουν λοιπόν δημιουργήσει αυτό αυτά τα γεγονότα, αυτές τις τρομοκριτικές ενέργειες, τεράστια πίεση στην ευαίσθητη ισορροπία συμβίωσης που υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει στην ε, Νιγηρία. Και η πρόκληση μας σήμερα είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δραστηριότητες των ομάδων αυτών έτσι ώστε να σταματήσουν να δολοφονούν, να σκοτώνουν αθώους και ταυτόχρονα να παγιώσουμε τις προσπάθειές μας για την οικοδόμηση πρωτοβουλειών οι οποίες θα οδηγήσουν στην ειρηνική συμβίωση όλων. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος με τον οποίο ε, οι χριστιανοί θα υπερισχύσουν στην Ιγυρία, ούτε οι μουσουλμάνοι θέλουμε να υπερισχύσουν στην Ιγυρία, είμαστε καταδικασμένοι, αφού ούτε ένας, ούτε άλλος θα επικρατήσει 100% να συμβιώσουμε. Αλλά δεν είναι καταδίκη, είναι και μία θετική και καρποφόρα συμβίωση. Αυτό θέλουμε. Είμαστε ε, μέλη διαφορετικών δογμάτων, πιστεύουμε σε διαφορετική θρησκεία, διαφορετικά δόγματα, αλλά πρέπει να δεχθούμε ότι συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες και αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις που μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε. σε ορισμένε περιοχές του Βορρά, όπως μόλις πληροφορηθήκαμε, πολιτικοί ή πολιτικά πρόσωπα έχουν υπερβάλλει ε, στο να τονίζουν τις σκεφτικές μας διαφορές και έχουν κάθε υπερβολή εδρεώσει ένα νομικό σύστημα βάσει της Σαρία που κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών αντιτίθεται στις ε, θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος μας. που λέει ότι δεν υπάρχει επίσημη κρατική δηλαδή θρησκεία στην Ιγυρία. Και η διαβούλευση από αυτού συνεχίζεται. Η Μπόκου Χαράμ, σα είπα, αυτή η οργάνωση μας ξάφνισε όλους. Ξάφνισε και την κυβέρνηση Δύο χρόνια, πήρε, δύο χρόνια χρειάστηκε η κυβέρνηση για να βρει τρόπο να μετοπίσει αυτή την οργάνωση. Υπάρχουν άνθρωποι, ε, οπαδοί αυτής της οργάνωσης που ο μόνος τους στόχος και ο μόνος τους σκοπός είναι να δολοφονούν γυριανούς πολίτες. Μερικές φορές η αντίδραση του κράτους δεν ήταν τόσο αποτελεσματική ως ίσως θα θέλαμε και οι κατηγορίες του ότι αντιμετωπίστηκαν με σκληρά μέτρα μπορεί εν μέρη να είναι σωστές, να υπάρχει μια βάσιμη κατηγορία, βάσιμος λόγος. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε. Και χτες πριν φύγω μάθαμε ότι έγινε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ορισμένων από αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις που απήγα, χρησιμοποίησαν τους ε, ε, κατοίκους χωριού ως ε, ασπίδες προστασίας κατά των, της επίθεσης των κυβερνητικών δυνάμεων. Αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα, ως ομήρους δηλαδή ουσιαστικά. Όχι μόνο ως χριστιανικός ηγέτης, που ανησυχώ και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τα χτυπήματα τα οποία έχουν υποστεί, πιστοί και που έχουν απαχθεί και απομακρυνθεί από τον τόπο κατοικία τους, αλλά με πληγώνει και ως Νιγηριανό, διότι κάθε ζωή στην Νιγηρία για μένα έχει αξία, είναι πολύτιμη. μου ζήτησαν να ε, αναφέρω και τις απόψεις μου για τις ελπίδες του μέλλοντος. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία ενδεικτικά που μας επιτρέπουν να είμαστε θετικοί, να είμαστε αισιόδοξη αν κάνουμε τα σωστά πράγματα και καταβάλουμε τις σωστές προσπάθειες να μπορέσουμε να επαναφέρουμε μια σωστή ειρηνική διακυβέρνηση στη χώρα μου έτσι ώστε τα τεράστια, η τεράστια ανθρώπινη δύναμη αλλά και ο πλούτος της χώρας να μπορούν τελικά να χρησιμοποιηθούν σωστά, θετικά για την ανάπτυξη της χώρας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από ό,τι κάνουμε τώρα. Επίσης, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Όχι μόνο και, και, παρόλο που υπάρχουν διαφορές φιλετικές και θρησκευτικέ, αλλά μπορεί να γίνει, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι διαφορές και δεδομένου ότι μπορούμε τις διαφορές αυτές να τις χρησιμοποιήσουμε ως πηγές, ως καλές θετικές πηγές πρόοδου. Πιστεύω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενισχύει αυτό το διάλογο τον οποίο άρχισα εγώ με άλλες συσκευτικέ ομάδες ε, στη χώρα μου. Γενικά δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να σας συναντήσουμε στη χώρα μου, ίσως διότι η εντολή σας δεν ε, ε, καλύπτει και τη συγκεκριμένη εντολή διαβούλευσης με θρησκευτικέ με θρησκευτικές ομάδες. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, σώμα και πολλά κράτη έχουν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν υποστηρίξει τις προσπάθειές μας ε, και με οικονομικό τρόπο και με άλλους. Και αυτή η υποστήριξη και συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί και πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν ανοίγματα και προς άλλες ομάδες του πληθυσμού μας έτσι ώστε να, έρθουμε και, να έρθουν και οι δύο πλευρές σε, επαφή σε καλύτερη συνεργασία να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη και έτσι να μπορέσουμε να εδρώσουμε, εν πάση περιπτώσει, μια ειρηνική συμβίωση σε αυτή την ωραία χώρα, την Ιγυρία. Θα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις ε, και θα μπορούσα να συνεχίσω επειδή ώρες για τη χώρα μου. Ε, έχετε την ευχή μου όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέντε αγωγητές έχω. Μπέλντερ πρώτος έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ισορροπημένη παρουσία σας εδώ. Και ευχαριστούμε που μας εξηγήσετε όλα αυτά στο Κοινοβούλιο. Είναι σύμπτωση αυτό, αλλά χτε με τον συνάδελφο κύριο Ντότζ ε, δεχθήκαμε ορισμένα θύματα της βίας από την Βόρεια Νιγηρία. Χθες είχαν έρθει στο Κοινοβούλιο. Μας έδειξε ένα φιλμ με, τις, με την κατάσταση στην χώρα ε, με εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες νεκρών από ε, ως θυμάτων του Μπόκο Χαράμ. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ είμαι προτεστάντης. Στη χώρα μου η Εκκλησία παρακολουθεί εκ του σύνεγγης της εξελίξεις στην Ιγυρία. Θέλω να θέσω μια σειρά ερωτημάτων, να μου επιτρέπετε. Μετά από αυτά που είδα χτες, για την ε, δίωξη των χριστιανών στην βορειοανατολική Νιγηρία. Μιλήσατε για δύο λέξεις που πλήττουν τη χώρα. Διαφθορά, έλλειψη ασφάλειας, ατιμορρησία. Η εικόνα που είχαμε και χθε στην ακρόαση είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ατιμορρησία κατά των δραστών αυτών των θρησκευτικού χαρακτήρα επιθέσεων. Εσείς ως υπερασπιστής του κλήρου και της Εκκλησίας στην Ιγυρία έχετε την πολιτική επίδραση και επιρροή στο κράτος για να χτυπήσετε αυτή τη βία που, βασιλεύει στη βορειοανατολική Νιγηρία. Γιατί, επαναλαμβάνω, Υπάρχει τεράστια ατιμορρυσία Και όταν συλλαμβάνονται οι δράστες, απελευθερώνονται αμέσω. Χτες οι παρευρισκόμενοι που ήταν καλά ενημερωμένοι μας είπαν ότι οι ακτιβιστές του Μπόκο Χαράμ έχουν παρισφρήσει και μέσα στο μηχανισμό του κράτους. Όταν είναι μέσα στο κράτος οι, οι τρομοκράτες, πώς μπορείς να χτυπήσεις την τρομοκρατία. Τι κάνετε λοιπόν, τι προσπαθείτε να κάνετε για να επηρεάσετε το κράτος τόσο ώστε να εμποδίσει αυτή την ε, ξέφρενη βία. Κατόπιν υπάρχει ένα, υπάρχει κά, υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο με, που προτάθηκε από 26 προσωπικότητες να δοθεί αμνηστία στο Μπόκο Χαράμ. Ε, αν γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά τι να σας πω, καλή επιτυχία θα σας έλεγα. Ο κύριος Κάλαμ. Σεβασμιότατε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που μας δώσετε για την κατάσταση στην Ιγυρία. Νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε το τραγικό γεγονός ότι τα προηγούμενα τρία χρόνια, 30 χρόνια, πολλοί δολοφονήθηκαν για θρησκευτικού λόγου. του τελευταίου χρόνου οι στατιστικέ μόνο είναι εντυπωσιακέ. Τον Απρίλιο 38 άτομα σκοτώθηκαν στην Καντούνα. Στι 29 Οκτωβρίου γύρω στα 50 άτομα δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας ενώ τραυματίστηκαν εκατοντάδε. Από ό,τι φαίνεται σε ένα χρόνο στην Ιγυρία υπάρχουν δεκάδες τέτοιες, ε, δεκάδες φαγές σαν αυτές που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη Βοστόνη, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για αυτές. Εξαιρετικά ανησυχητικό λοιπόν. Για τον Μπόκο Χαράμ. Το Μπόκο Χαράμ δραστηριοποιείται πια εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Ποιος τους υποστηρίζει. Πώς έχουν αποκτήσει αυτή την επίδραση που έχουν. Και τους επιτρέπει αυτή την θρησκευτική ή πολιτιστική εκαθάριση που, ε, που, εκαθάριση που εφαρμόζουν. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών. Μιλήσατε για την ε, διαφθορά και ένα γενικευμένο κλίμα ατιμορρησίας. Η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε να επηρεάσουμε, τι μπορούμε μαζί να κάνουμε για να επιβάλλουμε τη βελτίωση του κράτους δικαίου στην Νιγηρία και τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου που ήρθατε και μαρτυρήσατε για την πολύ περίπλοκη και δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην χώρα σας. Ερωτήσεις. Τον Μπόκο Χάραμ. Νομίζετε ότι είναι καθαρά ηθαγενής ομάδα αυτή. Και όπως ο Μάικλ Κέλαμ, ρωτώ και εγώ, Ποιο του υποστηρίζει, λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση απ' έξω, ξέρετε από ποιον. Αυτοί ισχυρίζονται ότι έχουν κάποιες διασυνδέσεις με την Αλκάιντα και ότι είναι ένα είδος ντόπιων αντιπροσώπων της. Εσείς γνωρίζετε για κάποια διασύνδεση με κάποια άλλη χώρα κάπου αλλού και αν δέχονται κυρίως χρηματοδοτική υποστήριξη και συνδέονται κατά ιονδήποτε τρόπο με άλλες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας όπως ίσως ναρκωτικά, λαθρεμπόριο, σωματεμπορία, ε, εμπόριο όπλων, έτσι ώστε να συλλέγουν χρήματα. Και η άλλη ερώτηση. Με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί ορθά επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει στην χώρα σας Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγείρει την φωνή της έτσι ώστε να ζητήσει από τις αρχές της χώρας σας να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους. Η Νιγηρία είναι εταίρος στους ΑΚΕ και δεσμεύεται από την Συμφωνία Κοτονού. Στέλνει και δυνάμεις της ε, μαζί με δυνάμεις της Αφρικανικής Ενώσεως και σε άλλες χώρες. Μήπως πρέπει λοιπόν, όπως είπα, να γύρουμε τη φωνή μας, μήπως είναι θέμα να συνεργαστούμε πραγματικά έτσι ώστε να φτιάξουμε το δυναμικό εκείνο που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά ή η ατιμορρησία των κυβερνητικών στελεχών ή υπάρχει κάποιο επίπεδο πολιτικής επιρροής που ίσως δεν έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σα υποβάλλω την ερώτηση αυτή διότι νομίζω ότι η κατάσταση που περιγράφεται απαντά και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ιγυρία. Σα ευχαριστώ. Σιμάνσκι από την ε, ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Σας ευχαριστώ εξοχότατε. Λαμβάνουμε πολλές πληροφορίες εδώ και πολλά χρόνια από την Ιγυρία, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τι προσωπικέ μαρτυρίε και εμπειρίες και ελπίζω ότι θα μας προσφέρετε κίνητρο και σε εμά και στα θεσμικά μας όργανα να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο στο τμήμα εκείνο του κόσμου που ε, γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλές και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Η θρησκευτική ελευθερία βέβαια έχει και την ατομική πτυχή γιατί είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα παίζει όμως και ζωτικό ρόλο για μια ειρηνική συνύπαρξη εν ειρήνη σε πολλά μέρη του κόσμου και βεβαίω και στην Ιγυρία. Θα ήθελα να σας ερωτήσω σχετικά με την ανταπόκριση σε αυτή την κατάσταση όχι μόνο από τις χριστιανικές κοινότητες που διώκονται στην Ιγυρία αλλά και από τις Ισλαμικές εκείνες κοινότητες που ασφαλώς δεν κυριαρχούνται ακόμη από αυτές τις ριζοσπαστικές μειονότητες ή μειοψηφίες που αποτελούν την αιτία των προβλημάτων για την ώρα. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν φόρα, υπάρχει βήμα όπου να μπορεί να συζητηθεί η βία που ασκείται στο όνομα των θρησκειών και για τις δύο κοινότητες, χριστιανική και μουσουλμανική. Και δεύτερη ερώτηση, παρόμοια όπως και άλλων ευρωβουλευτών, εσείς ως εκπρόσωπος της κοινωνικής πτυχής της Νιγηρίας. Τι αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και στο προσεχές μέλλον. Τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει σε αποκατάσταση της ειρήνης και σε μια ειρηνική συνύπαρξη στο προσεχές μέλλον στην Ιγυρία. Μπίσελτ. Ευχαριστώ ε, για την μαρτυρία σας στην, ε, για την κατάσταση. Μιλήσατε και για την ιδιαίτερη μοίρα των γυναικών ιδίως στο βόρειο μέρος της χώρας. Δύο ερωτήσεις. Εσείς θεωρείτε ότι συνδέεται η πρόοδος αυτή που κάνουν οι τρομοκρατικές ομάδες στο βορρά της χώρας με την φτώχεια. Βλέπουμε συχνά τις τρομοκρατικές αυτές ομάδες να ευημερούν ε, πάνω σε έδαφος φτώχειας. Διότι προσφέρουν κάποια κοινωνική ευημερία στις ε, φτωχές αυτές ομάδες, προσελκύουν δε έτσι τους νέους και τους πιθαναγκάζουν μετά να προβαίνουν σε τρομοκρατικές ενέργειες. Ανταποκρίνεται αυτό στην κατάσταση στην Ιγυρία. Βεβαίως η Νιγηρία είναι πετρελοπαραγωγός χώρα. Έχει σημαντικές πετρελαϊκές πηγές. Συνδέεται αυτός ο πετρελαϊκός πλούτος και η άνηση κατανομή του με την εμφάνιση αυτών των τρομοκρατικών ομάδων ή δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεγονότα. Εν τέλει δε, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοί μου, τι, τι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε στη δική σας, στον δικό σας αγώνα για μια λύση σε αυτό το δράμα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νιγηρία. Μενέντες Δελβάγε. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Γνωρίζετε καλά ότι το Ισλάμ γεννήθηκε έξι αιώνες μετά το χριστιανισμό. Και ο χριστιανισμός, όπως ξέρετε, είχε και αυτός εποχές φρίκης πριν από ευτυχώς πολλούς αιώνες. Φρικτές εποχές που θα έπρεπε να είχαν την ίδια καταδίκη και απόρριψη όποιες, όπως και ορισμένε ε, ε, φονταμενταλιστικές ε, ισλαμικές θέσεις τώρα. Κατά την άποψή μου και πιστεύω ότι και συμφωνείτε, κάθε είδους φανατισμός, ε, μουσουλμανικός, χριστιανικός ή εβραϊκός πρέπει να καταπολεμηθεί. Επίσης γνωρίζετε ότι δεν έχουν την ίδια κατάσταση ευτυχώς οι περισσότερες μουσουλμανικές χώρες, ούτε την ίδια στάση όπως αυτή που βλέπουμε στην Ιγυρία. Γνωρίζετε επίσης ότι η Ινδονησία για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε, η μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, είναι ευτυχώς η ακριβώς αντίθετη περίπτωση με της Νιγηρίας. Ρωτώ λοιπόν συγκεκριμένα στην οργάνωση της Ισλαμικής διάσκεψης υπάρχουν χώρες που χαίρονται για αυτά που συμβαίνουν στην Ιγυρία. Και η ερώτησή μου είναι, εσείς ως χριστιανικές κοινότητες στην Ιγυρία εξετάζετε το ενδεχόμενο να στραφείτε σε φορείς όπως η Οργάνωση Ισλαμικής Διάσκεψης για να διαμαρτυρηθείτε, να παρουσιάσετε τις θέσεις, να υποστηρίξετε τα επιχειρήματά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, να προσθέσω δύο σύντομες ερωτήσεις σε αυτές των συναδέλφων. Πρώτον, την πιθανή ύπαρξη ισχυρών εκτεταμένων αντιδράσεων στην Ιγυρία από το λεγόμενο μετριοπαθές Ισλάμ. Υπήρξαν θέσεις ισχυρές θέσεις καταδίκης του εξτρεμισμού και υποστήριξη των χριστιανικών κοινότητων της Ιγυρίας. Δεύτερον, το Μπόκο Χαράμ εδώ και πολύ καιρό κάνει επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας. Γι' αυτό χρειάζεται και εκπαίδευση και όπλη και, και υλικό για να διεξάγει τις, τις δραστηριότητες του αυτές. Αναφέρθηκε από συναδέλφους το ενδεχόμενο να δίδεται αυτή η χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές. Ρωτώ, μέσα στην Ιγυρία υπάρχει υποστήριξη, εκτεταμένη και σημαντική υποστήριξη προς τον εξτρεμισμό αυτό που και οι εκκλησίες που σκοτώνει κόσμο που αφαιρεί δηλαδή από τους πολίτες το δικαίωμα να ασκήσουν ένα βασικό, ένα βασικό δικαίωμα. Τέταρτο ερώτημα. Η σαρία, η θέσπιση σαρία δεν δημιουργεί de facto δύο διαφορετικές κατηγορίες πολιτών εφόσον οι νόμοι που εφαρμόζονται βάσει τη σαρία δεν είναι νόμοι που ισχύουν, ε, που εφαρμόζονται για την υπόλοιπη ένωμη τάξη της Νιγηρίας. Δημιουργούνται δηλαδή διαφορετικές κατηγορίες πολιτητών που εν τέλει θα μπορούσαν να ε, σπάσουν στα δύο τη χώρα. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε. Ευχαριστώ. Ρώτησα τον πρόεδρο πόση ώρα έχω να απαντήσω όλες αυτές τις πολύ σοβαρές και ε, θαυμάσιες ερωτήσεις. Βέβαια, πολλές ερωτήσεις επικαλύπτονται και σε 10 λεπτά θα μπορέσω ίσως να απαντήσω στις μισές. Ε, αλλά θα δούμε, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Καταρχάς, αλληλεγγύη, το ερώτηση για την αλληλεγγύη προς τα θύματα όλοι είμαστε θύματα. Ε, όταν διώκονται οι χριστιανοί δεν είναι ότι εξαιρείται η Ρώμα Καθολική Εκκλησία. Βεβαίω οι εκκλησίε μα είναι πολύ ορατέ, έχουν μια ισχυρή ε, παρουσία στι μεγάλε ε, πόλει και βεβαίω μα ανησυχούν πάρα πολύ αυτά τα σήματα. Δεν ξέρω ποια ομάδα ήταν αυτή που ήρθε χτες, αλλά το γεγονός είναι ότι υπάρχει ατιμορρησία. Υπάρχει ατιμορρησία στη χώρα μας. Και υπάρχει αυτή η προσέγγιση της ατιμορρητίας η οποία δίνει και την αυτοπεποίθηση στους ε, δράστες και, εκτελούν αυτές τις ε, πράξεις, τις ε, αποτρόπες πράξεις, ε, διότι πιστεύουν ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται σωστή δημοκρατική διακυβέρνηση, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι απλώς ε, υποσχέσεις χωρίς ουσία, αλλά εφαρμόζονται και ισχύουν στην καθημερινή ζωή. Ορισμένα μέλη με ρώτησαν τι μπορώ να κάνω εγώ ως ε, Ρωμακαθολικός ηγέτης και εάν ως καρδινάλιος έχω κάποια πολιτική επιρροή στην κυβέρνηση. Δεν έχω συγκεκριμένη πολιτική επίδραση, ούτε σχετίζομαι με πολιτικό κόμμα. Η μόνη πολιτική μου ισχύς είναι η δύναμη των μηνυμάτων μου. Οι, τα, τα, τα, οι δημόσιες ομιλίες μου στις συγκεντρώσεις, όπου εκφράζω τις απόψεις μου. Ε, πιστεύω ότι εκφράζω ρητά τις αρχές τις οποίες πιστεύω. Καλή διακυβέρνηση, ειλικρίνεια των πολιτικών ε, αρχηγών, φροντίδα ε, του πληθυσμού, φροντίδα για την δρέωση του κοινού ωφέλους για όλους, όλα αυτά τα καλά θέματα, τα καλά σημεία τα οποία τονίζω δύο από τα μέλη της κυβέρνησης είναι και πιστοί της εκκλησίας μου. Δεν ξέρω όμως εάν στα πολιτικά τους καθήκοντα ε, ενεργούν διαφορετικά από ότι ε, εγώ κηρύττω ή όχι, δηλαδή αν ακολουθούν τα κηρύγματά μου ή όχι. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίζω τα κηρύγματά μου. Η χώρα μου έχει δυνατή θρησκευτική ισχύ. Η, καθολική είναι 20%, 20%. Ακόμα και αν όλοι οι καθολικοί ακολουθούσαν τα κηρύγματά του, παραμένει το υπόλοιπο 80% της Νιγηρίας. Και τι κάνει το, ό, όλοι, αυτοί οι θάνατοι και οι δολοφονίες των τελευταίων ετών αποτελούν ντροπή για τη χώρα μου. Ορισμένες από αυτές τις, ε, τους θανάτους σημειώθηκαν για θρησκευτικού λόγους. άλλοι όμως πέθαναν από άλλες αιτίες. Τώρα, το Μπόκου Χαράμ ε, και η οργάνωση. Η κυβέρνηση πολλές φορές μας λέει ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά από ό,τι ξέρω εγώ δεν νομίζω ότι η οργάνωση αυτή έχει ε, ε, πάρα πολλά χρήματα και ότι κάνουν εισαγωγή ατελείωτων ποσοτήτων όπλων και ότι, ότι έχουν ας πούμε τεράστιες πηγές ε, και ότι όλα τα όπλα τα οποία περίζεψαν μετά την πτώση του κατάφη στη Λιβύη έχουν έρθει σε εμά, έχουν εισαχθεί στην Νιγηρία. Το θέμα είναι ότι ορισμένα από αυτά τα όπλα, ναι, προέρχονται από τις πηγές αυτές, αλλά μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές ε, επιδράμουν, επιτίθενται κατά αστυνομικών τμήματων και παίρνουν τα όπλα από εκεί. Χρησιμοποιούν δηλαδή εσωτερικές πηγές για την εξέβρεση των όπλων με την ευκαιρία αυτή θέλω να μιλήσω και για τη μουσουλμανική κοινότητα στην Ιγυρία. Στην αρχή οι, οι μουσουλμανικές κοινότητες αποκήρυταν την Μπόκου Χαράμ και έλεγα ότι αυτή η ομάδα η οποία θανατώνει εκτελεί μουσουλμάνους είναι κατά ε, του ε, ε, Ισλάμ δεν είναι γνήσιοι Ισλαμιστές είναι προδότες και όλοι αυτοί οι αυτοκτονοί ευωβιστές που αυτοκτονούν απαγορεύονται από το Ισλάμ αλλά εγώ πήγα και είπα ότι δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι είναι, είναι Ισλαμιστές, είναι μουσουλμάνοι και δεν μπορείτε να αρνηθείτε την ύπαρξή τους. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους να πλησιάσουμε την οργάνωση αυτή. Εκεί ακριβώς ακούστηκε και το θέμα της αμνηστίας. Ε, είπαμε κάποια στιγμή για αμνηστία, για να ενσαρρύνουμε ορισμένους από τους οπαδούς ε, της οργάνωσης που είχαν κουραστεί, είχαν αποτροπιαστεί τέλο πάντων από τις ε, τρομοκρατικές δράσεις και προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια διέξοδο προς τη συμφιλίωση. Η κυβέρνηση δέχτηκε θεωρητική να κάνει αυτή την προσπάθεια, να, να, να, να ρίξει αυτό το γάντι. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, τι καλό θα βγει, αν θα βγει. Αν θα σταματήσουν οι σκοτομοί, τότε μπορούμε να τους συγχωρήσουμε και να δώσουμε αμνηστία αν έχουν σταματήσει οι σκοτομοί και οι δολοφονίες για τα εγκλήματα δηλαδή που έχουν διαπράξει να δοθεί αμνηστία. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει σημειωθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα και ε, πολλοί από τους οπαδούς της οργάνωσης ε, λένε ότι δεν χρειάζονται την αμνηστία ούτε τους ενδιαφέρει διότι τα εγκλήματά τους δεν είναι εγκλήματα αλλά δικαιολογούνται. Επίσης είμαι ευτυχής που άκουσα ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι ε, ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και όπου δεν ε, επιτρέπεται η ανεξιθρησκεία υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώς. Το αυτό πιστεύω και εγώ. Τώρα τι περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς αυτό. Όπου υπάρχει έλλειψη θρησκευτικής ελευθερίας τότε θα πρέπει όσοι πιστεύουν να κράβονται και διακηρύσουν συνέχεια τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ακουστεί η φωνή τους έντονα και να πούν ότι αυτό είναι παράνομο και παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. πολλοί, πολλοί πιστεύουν και λένε ότι τα σκεφτικά δικαιώματα και η θρησκευτική ελευθερία δεν ανήκουν σε, στα, στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν εμπίπτουν σε αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Κάθε έθνος, κάθε κράτος είναι υπόλογο για τη συμπεριφορά των πολιτών. Και στην ε, Δεύτερη Αφρικανική Σύνοδο το είπαμε αυτό σαφέστατα στα, στα συμπεράσματα που δημοσιεύσαμε ότι μια κυβέρνηση η οποία δεν επιτρέπει την ελευθερία του πιστεύω, την θρησκευτική ελευθερία στους πολίτες της παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που σημαίνει ότι ορισμένες χώρες που λένε ότι είναι οι χριστιανικές, ή μουσουλμανικές και δεν επιτρέπουν την ελεύθερη έκφραση της πίστης στους άλλους που δεν είναι, ε, θα πρέπει να ε, καταδικάσετε. Τώρα, σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και ε, φτώχειας. Ναι, ίσως, αλλά η φτώχεια από μόνη της δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί στην Ιγυρία που δεν είναι ούτε τρομοκράτες, ούτε αλήτες. Όπου έχουμε φτώχεια, αυτή οφείλεται κυρίως στην ε, άνηση, εντελώς άνηση κατανομή του εθνικού πλούτου. Όταν υπάρχει αυτή η ανισοκατανομή δημιουργείται και απελπισία, δημιουργείται και φτώχεια μεγάλη και βεβαίως πολλοί από αυτούς που υποφέρουν ε, είναι διαθέσιμοι να ακούσουν ή να ακολουθήσουν διάφορους κακούς σκοπούς. Και υπάρχουν ε, υπάρχει τρόπος η κυβέρνηση να βρει τρόπους να καταπολεμήσει ε, τα φαινόμενα αυτά της τρομοκρατίας όταν έχουν σχέση με την διακίνηση ναρκωτικών. Άκουσα ότι μία ομάδα στο Μάλι έχει επιβεβαιωθεί ότι διακίνει ναρκωτικά. Ε, έχω την υποψία, αλλά όχι τη βεβαιότητα, ότι χρησιμοποιούν ε, των λαθρεμπόριων ναρκωτικών ως πηγή πλούτου, ας πούμε πηγή χρηματοδότησης. Το παράδειγμα της Ινδονησίας είναι ενδιαφέρον. Τα μηνύματα από την Ινδονησία τα τελευταία δύο χρόνια είναι ε, θετικά, αισιόδοξα. Είναι μια χώρα όπου οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι όχι μόνο ζουν ειρηνικά, συμβιώνουν ειρηνικά, αλλά σέβεται και μία κοινότητα την άλλη. Στην Νιγηρία δεν ε, απαιτώ, απαιτώ την ανεξιδρυσκεία, απαιτώ την ελευθερία πίστης, την ελευθερία άσκησης της θρησκείας μου και 80 εκατομμύρια χριστιανοί και 80 εκατομμύρια μουσουλμάνοι που είναι τεράστιος αριθμός πληθυσμού, έχουμε συμβιώσει, έχουμε πετύχει στη συμβίωση. Δεν νομίζω ότι μία μικρή τρομοκρατική και αρχαία ομάδα μπορεί να διαγράψει όλα τα καλά, όλες τις επιτυχίες που έχουμε σημειώσει μέχρι τώρα. Όσον αφορά τώρα τους μετριοπαθείς μουσουλμάνους, εγώ δεν θέλω να με χαρακτηρίσουν μετριοπαθή χριστιανό. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στην ειρήνη, που έχουν σωστή θέληση, ε, που, που είναι εναντίον του Μπόκου Χαράμ και πολλές φορές ε, ε, οι άνθρωποι αυτοί που εκφράζονται υπέρ της ειρήνης και της συμβίωσης έχουν δεχτεί επιθέσεις από την Μποκοχαράμ, αποτελούν στόχο. Δεν είναι λοιπόν σωστό ότι όλοι κυνηγούν και επιτίθενται κατά των χριστιανών. Ορισμένοι χριστιανοί βεβαίως αισθάνονται ε, διωγμένοι και υποπίεση, αλλά εκτός από την Μπόκου Χαράμ, εκτός δηλαδή της εμβέλειας του Μπόκου υπάρχουν, υπάρχει και αυτή η πίστη. an opinion that Άποψή μου είναι ότι η Σαρία ξεκίνησε σε κάποιες πολιτείες από τους πολιτικούς, όχι από την θρησκευτική ηγεσία, με βάση μια θρησκευτική ατζέντα που δεν ήταν η ατζέντα της θρησκείας. Εάν δεν αλλάξει αυτό, θα υπά, συνεχίσουν να υπάρχουν κακές σχέσεις μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Κοίταζα τις ε, ερωτήσει: Τι μπορεί να κάνει περισσότερο η Ένωση. Φωνάξτε. Δεν ξέρω αν δεν φωνάζετε, αλλά αν δεν φωνάζετε φωνάξτε. Μπορεί να υπάρχουν διπλωματικοί τρόποι να τα πείτε, πείτε τα όμως. Ε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε περισσότερο στην ε, καλή διακυβέρνηση. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε, να, να, να επιβάλλετε τις θέσεις στους πολιτικούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε εκλογές και όταν έχετε σαφείς ενδείξεις μαζικής νοθείας κάποιοι από εσά που είναι παρατηρητές ε, και πιστεύετε ότι δεν έγιναν σωστά οι εκλογές. Αρχίζουν οι χαρές, οι ενθουσιασμοί των νικητών και πριν αλέκτρο λαλήσει τρέχουν τα συγχαρητήρια από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη. Αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Η μόνη εξαίρεση είναι η στρατιωτική, η ανάλυση δικτατορία. Μην ξεχνάτε ότι, κάποια, ότι ξεχάσαμε τώρα ότι υπήρχαν ε, στο παρελθόν ε, στρατιωτικοί δικτάτορες, τους οποίους κα, καταδικάζεται. Πιστεύω ότι όταν οι δικτάτορες οι κλέφτες του εθνικού πλούτου δεν αντιμετωπίζονται με σεβασμό στο εξωτερικό, θα είναι λιγότερο ελκυστικό να αναλάβεις την εξουσία και να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν λέω ότι η χώρα μου είναι έτσι, αλλά έχουμε κάποια στοιχεία. Και αυτό με οδηγεί στην πολιτική επίδραση. Πόσο πολιτική επιρροή έχει ένα κράτος ένα άλλο κράτος. Και πρέπει να έχει πριν γίνει παρέμβαση στα εσωτερικά. Άποψή μου είναι ότι οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να μας δώσετε, τόσο καλύτερα. Μιλώ ελεύθερα στους, ε, στο πίμνιό μου και τους λέω ποιο πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα του έθνους μας και το λέω και σε εσά τώρα, να είχαμε μια μεγαλή η φωνή, ούτως ώστε να επηρεάσουμε αυτούς που έχουν ή θέλουν την εξουσία για να τους επηρεάσουμε ούτως ώστε να κάνουν καλύτερη δουλειά προς όφελος όλων. Μια καλύτερη διακυβέρνηση της χώρας θα οδηγήσει σε μείωση της δίωξης και των χριστιανών. Ευχαριστώ. Είπατε πολλά σε λίγο χρόνο.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 as a souvenir. Uh, next. Ακολουθεί τώρα η σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύμπραξης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και Μαλαισίας. Με εισηγητή τον κύριο Μενέντες Τελβάγε, που είναι παρόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για την συμφωνία αυτή η αρμόδια της ουσίας είναι η Επιτροπή Εξωτερικών. Η δε ίντα είναι αρμόδια για γνωμοδότηση. Έχει προχωρήσει η συμφωνία αυτή, αλλά έχει τώρα ανασταλεί η διαπραγμάτευση λόγω των εκλογών στη Μαλαισία στις 5 Μαΐου. Γίνονται ανταλλαγές απόψεων και σήμερα ανταλλαγή απόψεων μάλλον η δε τελική προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών θα είναι η 7η Μαΐου το μεσημέρι. Από πλευράς μου αυτά και δίνω αμέσω τον λόγο στον εισηγητή κύριο Εμίλιο Μενέντε Τιλβάρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το σχέδιο περιλαμβάνει μια σειρά συστάσεων για τις διαπραγματεύσεις ε, τη Συμφωνία Σύνδεσης και συνεργασία που αναφέρεται. Στο ίδιο κείμενο περιλαμβάνω τέσσερις ε, τομείς σημαντικούς για τις δύο πλευρές Ένωση και Μαλισσία τις διαπραγματεύσεις αυτές καθευτές, τον πολιτικό διάλογο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αμελαιώδεις ελευθερίες και την οικονομική, πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης, θεωρώ θετικό να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ιδίως τη Μαλαισία στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάντα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγει η Ένωση με τις άλλες, με άλλες πέντε χώρες του ΑΣΕΑΝ. Για το δεύτερο θέμα, τον πολιτικό διάλογο, είναι σκόπιμο να επενέσουμε τον υψηλό βαθμό υποπεριφερειακή συνεργασία στις Μαλαισίας μέσω σημαντικών πρωτοβουλειών ασφάλειας της θάλασσας στην ε, περιοχή. Ένα εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα σε αυτή την ε, περιοχή, όπως ξέρετε, καθώς και την υποστήριξη της Μαλαισίας της ε, προσπάθειες καταπολέμησης της πειρατείας στην ακτή της Ομαλίας, κάπου σημείο στο οποίο εμπλέκεται και η Ένωση. Ταυτόχρονα αναγνωρίζω τις προσπάθειες των αρχών της χώρας για την αξιέπαινη ε, προσπάθειά τους για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, τα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως το δημοκρατία ξέπλυμα χρήματος κλπ. Διαφοροποιώ, υπογραμμίζω επίσης την εξαιρετική περίοδο μακράς σταθερότητας μέχρι τις εκλογές του 8 στην χώρα και ζητώ από τις ε, αρχές ε, που, που θα βγουν από τις εκλογές του Μαΐου του 2013 να δώσουν σημασία στην πολιτική και εθνοτική ένταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η χώρα και προτείνω να προχωρήσουμε η υποχρέωση είναι προ την ενίσχυση ενό ισχυρού διαλόγου με την ε, αντιπολίτευση της διάφορε εθνοτικές ομάδε, ε, να υιοθετηθούν μέτρα καταπολέμηση τη διαφθορά και να συνεχιστούν οι οικονομικέ και πολιτικέ μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι εμελίδε ελευθερία, καλωσορίζω την δέσμευση τη κυβέρνηση να καταργήσει, να αντικαταστήσει την ε, θανατική ποινή με τα ισόβια δεσμά, όπως αναγγέλθηκε το 2009 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Άλλο σημαντικό μέτρο ήταν η αντικατάσταση του νόμου εσωτερικής ασφάλειας από το νόμο για την, τα εγκλήματα ασφάλειας που περιορίζει την maximum περίοδο κράτησης ενός πολίτη χωρίς κατηγορία ή δίκη. Παρά τα αυτά ο, ο νόμος αυτός έχει ακόμα πολλά κενά σε ό,τι αφορά το καθεστώς των ε, εφέσεων και την στέρηση της ελευθερίας. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό του τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρώ σκόπιμο να απευθυνθώ, να απευθύνω έκκληση προς την κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλίσει τα συνταγματικά δικαιώματα σε όλους τους πολίτες, όπως και είδαμε τι έγινε στην Ιγυρία τώρα, όπως την ελευθερία έκφρασης ε, της θρησκευτική λατρείας και την ε, ενίσχυση της ανεκτικότητας και του διαθρησκιακού διαλόγου που δεν είναι πρόβλημα μόνο της Νιγηρίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων στη Μαλαισία συγκεκριμένα και την πολιτική και δικαστική παρέμβαση που δημιουργεί κίνδυνο αποδυνάμωσης του καθεστώτος των γλωσσικών εθήμων που είναι μια εκτεταμένη κατάσταση στη χώρα. Επιπλέον, στον τομέα της επιστημονικής ε, και πολιτιστικής συνεργασίας θέλω να συγχαρώ τις αρχές της χώρας για την βαθιά δέσμευσή τους υπέρ της προώθησης της ενεργειακής ε, αποτελεσματικότητας, της χρήσης των, ε, και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολλές άλλες πράσινες ε, πρωτοβουλίες. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να παρατείνω άλλο την παρέμβασή μου. Θα περάσουν ε, πολλά θέματα σε τροπολογίες. Απλά υπογραμμίζω ότι ε, η χώρα πρέπει να προχωρήσει στην ελευθερία πληροφορίας όπου υπήρξαν μεν βελτιώσει αλλά όχι επαρκείς. Κατά την άποψή μου επίσης η ελευθερία του συναθρίζεστε δεν είναι επαρκώ προστατευμένη, ιδίω στι αστικέ περιοχές. Ε, επιπλέον, είπαμε ότι καταργήθηκε η ποινή του, θα καταργηθεί η ποινή του θανάτου, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν οι σωματικέ τιμωρίε στην χώρα. Επίση, η Μαλαισία πρέπει να τηρήσει τα διεθνή στάνταρ εργασία κυρίω δε τι προδιαγραφέ του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασία με τι οποίε συμφωνούμε όλοι, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθε. Αυτό βέβαια αφορά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι κατεστημένες εκεί. Τέλος, να τονίσω ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τον οικολογικό τουρισμό. Η Μαλαισία έχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για να, για να γίνει ο τουρισμός αυτός ελκυστικός. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη της χώρας. Είπα ό,τι έπρεπε να πω πρόεδρε. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πρόεδρε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Λίζεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας στην ουσία με πρόλαβε και είπε όλα όσα θα ήθελα να πω κι εγώ. Πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ καλά η έκθεση. Η έκθεση είναι σχεδόν πλήρης αφού περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της κατάστασης στην Μαλαισία και βεβαίως τη συνεργασία μας με τη χώρα αυτή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σημασία της συνεργασίας μας με την Ασία και τις χώρες του Νότιου Ειρηνικού η σημασία λοιπόν αυτή θα αυξηθεί όπως θα αυξηθεί η σημασία της περιοχής αυτής του κόσμου. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η Μαλαισία συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που θα ενισχυθεί ο ρόλος τους στην περιοχή αυτή. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον κύριο Μινέντε Τιλβάγε που έθιξε ποικιλία θεμάτων που έχουν σχέση με τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή και ως αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής της Αρμόδιας Επιτροπής ήθελα να πω ότι η Μαλαισία είναι σημαντική για την σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή αυτή του κόσμου και συμμετέχει σε διάφορους οργανισμούς που επιδιώκουν τη διασφάλιση της ειρήνης. Τονίσατε επίσης ότι και εμείς υποστηριζόμαστε από τη Μαλαισία σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μέτρα για την καταπολέμηση της πειρατείας στην ε, ακτή της Σομαλίας. Η Μαλαισία θα παίξει αναμφίβολα σημαντικό ρόλο και στη νότια Κινέζικη θάλασσα. Και χαίρομαι που αφιερώνεται τόση προσοχή στο θέμα. Η Μαλαισία από τη σκοπιά μας βέβαια δεν είναι άψογη όσον αφορά τα συστήματά της. Σημειώνουμε ωστόσο με ικανοποίηση τις κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν στη χώρα αυτή. Ωστόσο, οφείλουμε να ζητήσουμε από τους εταίρους μας Μαλαίους να επιταχύνουν τις διαδικασίες αυτές, λαμβάνοντας εντονότερα, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, ελευθερία της ε, θρησκείας Ελευθερία συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και πάντως μπορείτε να αναμένετε την υποστήριξη της πολιτικής μου ομάδας. Εν τέλει δε θέλω να πω ότι θεωρώ σημαντικό η διακοινοβουλευτική συνεργασία που, που μάλλον η διακοινοβουλευτική συνεργασία επίσης βρίσκει χώρο στην έκθεσή σας. Η κυρία Γκόμες. Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να συγχαρώ τον κύριο Μενέντε Τελβάγε για την σε βάθος ε, μελέτη του θέματος και επικοδομητική εκθεσή του περιλαμβάνει πολλές θετικές συστάσεις για το Συμβούλιο Υπουργών και για την Κομισιόν στην διαπραγμάτευση της Συμφωνίας Συνεργασίας με τη Μαλαισία. Συμφωνώ ότι η Μαλαισία είναι σημαντικός εταίρος μεταξύ των ασιατικών χωρών και ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τις σχέσεις μαζί τους από κάθε άποψη, βεβαίω και περιλαμβάνω εδώ και την κοινοβουλευτική πτυχή. Συμφωνώ με τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες που τονίζει και ο εισηγητής, διότι παρά την ζωηρή συζήτηση που γίνεται στη Μαλαισία, Υπάρχουν ωστόσο ακόμη σημαντικές ανησυχίες, όπως για παράδειγμα η θανατική ποινή. Η πρότασή μου είναι για το θέμα της συνεργασίας στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, πλησίματος μαύρου χρήματος, διαφόρων σωματεμποριών κτλ. να περιλάβουμε και την πτυχή της καταπολέμησης του απόρριτου των φορολογικών παραδείσων. Κάτι που απασχολεί όλο και περισσότερο για την περιοχή αυτού του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει, αυξάνεται και γίνεται οικονομικά όλο και πιο σημαντικό. Η Μαλαισία θεωρώ με το Ισλαμικό σύστημα που διέπει την ζωή της μπορεί να μας προσφέρει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις πιο αρνητικές πτυχές αυτής της φυγής κεφαλαίων. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί και αυτός ο χώρος να αποδειχθεί σημαντικός για τη συνεργασία. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ που με καλέσατε στη συνάντηση αυτή. Είναι χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Είναι το ξεκίνημα της θητείας μου. Μόνο 1η Φεβρουαρίου ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Διαβάσαμε την έκθεση, πολύ ενδιαφέρουσα, πλήρης. Εξετάζουμε εκ του σύνεγγης της ε, συστάσεις. Όπως είπε και ο εισηγητής, ε, ο ρόλος της Μαλαισίας ε, είναι πολύ σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η συμφωνία είναι ένας καλός τρόπος να εμπλέξουμε να την αυξήσουμε τη συνεργασία σε μια σειρά θεμάτων παροτρύνοντας ε, τη χώρα να προχωρήσει παρατέρα και τούτο θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε σύντομα ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων και θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής για να κλείσει. Σύντομα. Πρώτον, ευχαριστώ τους συναδέλφους που μίλησαν για τα σχόλια που κάνατε. Ευχαριστώ. Κατά την άποψή μου, δεν είναι ότι είναι εξαιρετική η έκθεση, αλλά ότι υπάρχει συμφωνία επί γεγονότων συγκεκριμένων, σαφών, που απαιτούν λύσεις που συμμερίζονται και οι συνάδελφοι και εσείς, πρόεδρε, φαντάζομαι, διότι είναι βασικό αυτού. Ευχαριστώ την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τα σχόλιά του που συγχαίρω και για την πρόσφατη πρόσληψή του. Κλείνω λέγοντας ότι, όπως γνωρίζετε, Πρόεδρε, η προθεσμία για την υποβολή των τομπολογιών είναι 7 Μαΐου. Αυτά. Ευχαριστώ. και εγώ. Επόμενο θέμα. Τώρα, στην μερίσια διάταξη έχουμε την ανταλλαγή απόψεων με την Αν Τζένσεν, εισηγήτρια τη Επιτροπή προπολογισμών. για τον προπολογισμό το 2014. Ανταλλαγή απόψεων. Αυτό θα είναι μια πρώτη συζήτηση για τις προτεραιότητες ε, της ΑΦΕΤ πριν από την παρουσίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και αποτελούν τμήμα ε, των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων με το πολιετές ε, πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα αυτό βασίζεται και στο περσινό χρονοδιάγραμμα είναι μια πολύ καλή και εύκαιρη χρονική στιγμή να μας ενημερώσει η κυρία Τζένσεν και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω για την κατάσταση και να ακούσω τις δικές σας απόψεις είναι σημαντικό τμήμα των διαδικασιών του προϋπολογισμού να λαμβάνουμε τις απόψεις των ε, επιτροπών. Εμείς ψηφίσαμε ε, τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2014 το Μάρτιο στο Στρασβούργο και αν θυμόσαστε αυτό το ψήφισμα που υπερψηφίσαμε είχε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορούσε με το γεγονός ότι δεν έχουμε ένα πολιετές πλαίσιο αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε και τη νομική βάση. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ παράδοξη κατάσταση όπου όλο το πλαίσιο ε, του ετησίου προπολογισμού δεν υπάρχει. Δεύτερον, έλεγε το ψήφισμα ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε προβλήματα με το Συμβούλιο, που δεν είχε την θέληση να ορίσει επαρκής πιστώσης πληρωμών. Είναι τεχνικό μεν το θέμα. Οι πληρωμές από τη στιγμή που έχεις αναλάβει τη δέσμευση ε, πρέπει να γίνουν. Και ε, πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό από τη στιγμή που έχει εκδοθεί. Όμως ε, φαίνεται ότι το Συμβούλιο ερμηνεύει διαφορετικά τα πράγματα και όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι το πρόβλημα αυτό των πληρωμών γίνεται και πολιτικό πρόβλημα. Βέβαια, ε, είναι κυρίως πρόβλημα στην ε, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων, αλλά και στην ΑΦΕΤ νομίζω μπορεί να αποτελέσει ένα πρόβλημα διότι εμπίπτει στον τομέα της πολιτικής, των πολιτικών. Επίσης, το τρίτο θέμα είναι ότι αναφέραμε τις πολιτικές προτεραιότητες, την ανεργία των νέων και τη στρατηγική του 2020. Και βέβαια, αυτό ίσως δεν αφορά τόσο πολύ την ΑΦΕΤ, αλλά και εσείς έχετε ε, απόψεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη στη διαδικασία μας. Ε, αλλά το, το θέμα αυτό συνδέεται με τις διαβουλεύσεις του MMF, του πολιετούς πλαισίου, για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε τη νομική βάση για τα προγράμματα από το 2014 και πέρα. Και όλες οι επιτροπές τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν ακριβώς φόρμες για τον προϋπολογισμό. Έχουμε λάβει από την Κομισιόν και ελπίζω να έχει διατεθεί και σε εσά, αλλιώ θα σας το δώσω, μία μετάφραση από την Κομισιόν τη συμφωνία που έγινε το Φεβρουάριο μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, όπου αποφασίστηκε ένα πλαίσιο του προπολογισμού το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό πρότεινε η Κομισιόν και χαμηλότερο από αυτά που επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από αυτού τώρα διαπραγματευόμαστε. Η Κομισιόν άτυπα τώρα προσπάθησε να ερμηνεύσει αυτή τη συμφωνία και εάν ε, είδατε ε, τα αριθμητικά στοιχεία δεν θα είστε πολύ ευτυχείς. Είναι στοιχεία τα οποία είναι κατώτερα των επισημειών αυτής της Επιτροπής. Θα με ρωτήσετε τι ελπίδες μπορεί να έχουμε τώρα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των πολιετών, του πολιετούς πλαισίου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι την τελευταία φορά που έγιναν διαβουλεύσεις το Κοινοβούλιο κέρδισε 5 δις περισσότερα για 7 χρόνια. Ε, θα είναι λοιπόν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις για να πάρουμε περισσότερα χρήματα και θα συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ε, στην ευελιξία και στην, ε, στο να δαπανηθούν οι πληρωμές με καλύτερο τρόπο, επίσης σε έναν σαφή καθορισμό των προτεραιοτήτων και στην παρακολούθηση ε, των εφαρμογών, δηλαδή της ε, υλοποίησης ε, των καταβολών, των πληρωμών, που πηγαίνουν τα λεφτά, αν χρησιμοποιούνται σωστά κλπ. Παραδείγματο χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία έχει μια σωστή υλοποίηση των πληρωμών και είναι ένας από τους τομείς όπου θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε υψηλότερα κονδύλια. Αναμένουμε τέλος Μαΐου την πρόταση της Κομισιόν και ε, τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία, τα ποσά ε, θα βασίζονται στους δικούς τους υπολογισμούς και θα δούμε πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα ελπίζω να έχουμε βρει και μία λύση για το πολιετές πλαίσιο και τη νομική βάση. Χρησιμοποιήθηκε ε, και, και ένα άλλο μέσον, πιλωτικά προγράμματα ε, και το ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή σας. Και εδώ πρέπει να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες από τις Επιτροπές μέχρι το τέλος ε, του Μαΐου. Νομίζω έχει μας έχουν στείλει οδηγίες για το πώς θα διαμορφώσουμε τις 10 look through and see whether they find the ideas feasible uh, or whether by by programs that will already be. Πώς θα παρουσιάσουμε τις απαιτήσεις μας, τις προτάσεις μας για τα 10 και ε, τις γραμμές δηλαδή για τα προγράμματα που εμπίπτουν στα ΤΕΝ και ελπίζω για τον προϋπολογισμό 2014 ε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε εν μέρη τουλάχιστον και γι' αυτό σας έδωσα όλο αυτό το ιστορικό υπόβαθρο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αναμένουμε τον εισηγητή. Αλλά βέβαια είναι απόν για την ώρα. Αλλά άλλες ερωτήσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν. Μεγάλη επιτυχία κυρία Γένσεν. Θα διακόψουμε μέχρι τις 4.45 μέχρι ότου έρθει η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα. 4.45 ακριβώς. Ο πρόεδρος Μπροκ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Κριστίν, μην επηρεάζει πολύ τον συντονιστή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Χαριτολογεί ο πρόεδρος Μπροκ. Έχουμε κοντά μας τώρα την Επίτροπο κυρία Γεωργίευα, με την οποία θέλουμε να συνομιλήσουμε για θέματα Συρίας, της καταστάσεως εκεί, και βέβαια και το θέμα των προσφύγων σε Ιορδανία και Λίβανο. Υπάρχουν πολλοί στους δρόμους. Ακούσαμε και σήμερα για τους ε, επισκόπους, για τους αρχιεπισκόπους μάλλον, που απήχθησαν. Υπάρχουν νέα. Πιθανώς απήχθησαν από ανθρώπους της αντιπολίτευσης. Ήρθε και ο Υπουργό κ. Φαμπίου την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή μα, με, την οποία τον οποίο συζητήσαμε μάλλον την Συρία και την κατάσταση στι γειτονικέ χώρε. Το Μάλι επίση. Χιλιάδε άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Συρία από την αρχή των συγκρούσεων εκεί. και πάνω από 4 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι στην ίδια τη Συρία και οι ε, πρόσφυγες και στον Λίβανο και στην Ιορδανία αποτελούν ίδιο ανθρωπιστικό πρόβλημα αλλά και υπάρχει και κίνδυνος αποσταθεροποίησης των χωρών αυτών. Άρα είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις και βεβαίως και το βάρος που συνεπάγονται οι πρόσφυγες αυτοί για την Τουρκία που εμπλέκεται βεβαίως στη μεγαλύτερη, στην ευρύτερη αυτή ε, ε, ε, σε ευρύτερο αυτό θέμα και πρόβλημα. Το κόστος για, την στήριξη των προσφύγων ανέρχεται στο 3% το ΕΠ της χώρας. Είναι πολλά χρήματα. Όταν οι δικές μας χώρες μέλη θεωρούν ότι 1% να εισφέρουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υπερβολικά πολύ. Έτσι λοιπόν κυρία Επίτροπε, χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ για την διάθεσή σας να μας ενημερώσετε. Και για λόγους πολιτικούς αλλά και ανθρωπιστικούς είμαστε διατεθειμένες και διατεθειμένοι να ενισχύσουμε την προσπάθειά σας. Η κυρία Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πράγματι επίκαιρη η στιγμή να εστιάσουμε την προσοχή μας στη Συρία και στην γειτονιά της και να δούμε τι μπορεί να κάνει η διεθνής κοινότητα δοθέντος του πολιτικού αδιεξόδου που ακόμα δεν έχει ε, ξεπεραστεί. Ακούσαμε ισχυρή φωνή από την ανθρωπιστική κοινότητα με πέντε επικεφαλής ε, οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών που σε κοινή τους δήλωση είπαν φτάνει. Έχουμε φτάσει σε τόσο αυξημένο κίνδυνο στην Συρία και στις γειτονικέ της χώρες που σημαίνει πλέον αυξημένο κίνδυνο και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Σεις μιλήσατε για τα γεγονότα που όσο τρομερά κι αν είναι, ακόμα τρομερότερο είναι να εξετάσει κανείς τις ενδεχόμενες διαγραφόμενες τάσεις και στην Συρία και στην άμεση γειτονιά της. Θα σας δώσω τρία σημεία αναφοράς. Πρώτο, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι στην Συρία μέσα στους τελευταίους μήνες έχουν διπλασιαστεί από 2 σε 4,3 εκατομμύρια ανθρώπων ως σημείο αναφοράς στην κρίση της πρώην Ιουκοσλαβίας, στο σύνολό της, είχαμε οδηγηθεί σε 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους. Η αύξηση των, του αριθμού των προσφύγων. Χθε, μιλούσα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Εγώ παρακολουθώ τις μετρήσεις που κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη καθημερινά στην ιστοσελίδα των προσφύγων. χθε είχαν φτάσει στο 1.370.000 πρόσωπα. Όταν έφυγα να έρθω εδώ στο κοινοβούλιο σας, ξανακοίταξα και ο αριθμός έχει φτάσει στο 1.381.000 και πάνω, δηλαδή 11.000 αύξηση μέσα σε μια μέρα. Εάν οι προβολές του ΥΠΑ του αρμοστή των προσφύγων υλοποιηθούν μέχρι τέλους του έτους, θα έχουμε φτάσει στα 3,5 εκατομμύρια προσφύγων. Ένα εκατομμύριο στην Ιορδανία, ένα στον Λίβανο, ένα στην ε, ε, Τουρκία και το, και το υπόλοιπο στην Αίγυπτο και στο Ιράκ. Το σύνολο, επαναλαμβάνω, των προσφύγων από την κρίση της Ιουγκλαβίας ήταν 700.000 άτομα. Και το χειρότερο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι στο Ιράκ 2 εκατομμύρια. Και από Λίβανο και η Ορδανία, για τον Λίβανο και την Ορδανία, τέτοιου είδου αύξηση σημαίνει είναι ότι ο πληθυσμός τους θα αυξηθεί κατά 20-30%. Εδώ στην Ευρώπη ποια χώρα μας θα ήταν ικανή να δεχθεί να εποπτεύσει ε, αστυνομικά και να προσφέρει υπηρεσίες σε 20% παραπάνω πληθυσμό μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Άρα η κίνδυνη να ξεχυθεί αυτό και στις γειτονικές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήδη βλέπουμε επιτόπου στο Λίβανο αλλά και στην Ιορδανία κοινότητες που είχαν φανεί πολύ φιλόξενες στους Σύρους πρόσφυγες να γίνονται πιο αρνητικές και ο ιός της διακοινωτικής βίας να αρχίσει να είναι πιθανό να εξαπλώνεται με τρομακτικές συνέπειες για τις χώρες και για την ευρύτερη περιοχή. Επιθυμώ να θέσω δύο θέματα τώρα για την απαραίτητη δράση. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις των ΗΠΑ και οι μη κρατικοί οργανισμοί έχουν αυξήσει την παρουσία τους και έχουν διατεθεί πόροι επίσης οι οποίοι αυξάνονται. Όμως, λόγω της αυξανόμενης βίας όλο και μεγαλύτερο το χάσμα. Πάνω από 30 συνεργάτες ανθρωπιστικών οργανώσεων έχασαν τη ζωή τους. Πολύ περισσότεροι έχουν απαχθεί ή έχουν τραυματιστεί. Η ικανότητα προσφοράς ωστόσο είναι περιορισμένη και περιορίζεται και ακόμη περισσότερο λόγω παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και επομένως περιορίζεται ο χώρος για να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε. Το δεύτερο τώρα είναι η αντοχή των ίδιων των σύρων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι σύροι βοηθούσαν σύρους και ε, αυτή ήταν η προστασία κατά της κρίσης. Αυτή η ικανότητα των ανθρώπων προς αυτοβοήθεια μειώνεται σοβαρά. Θα σας δώσω έναν αριθμό που για μένα ε, ήταν ε, μια τρομερή έκπληξη. Στο Χαλέπι είχε 5.000 εγγεγραμμένους γιατρούς. Σήμερα έχουν μείνει 36. Ορισμένοι σκοτώθηκαν, άλλοι έφυγαν. Και αυτή είναι η εικόνα σε ολόκληρη τη Συρία. Είναι λοιπόν ένα τρομερά σημαντικό ηθικό θέμα η κινητοποίηση βοήθειας για τη Συρία και για τις γειτονικές της χώρες. Αλλά είναι και προς το δικό μας συμφέρον η κίνδυνη έκχυση των κινδύνων, αυτό το spillover, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερο θέμα. Πρέπει να παραγάγουμε μια νέα όθηση, ένα συνολικό πρόγραμμα για την στήριξη των σύρων αλλά και των γειτονικών χωρών. Εκεί απαιτείται η ηγετική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω ακόμα τρεις συγκεκριμένες συστάσεις δράσεων που μπορούμε να αναλάβουμε σε αυτή την πολύ δραματική κρίση. Κρίση που δεν με αφήνει να κοιμηθώ κύριε Μπρόκ Πρώτα, λόγω του πόνου και της δυστυχίας στη Συρία είναι απαραίτητο να πιέσουμε να ανοίξει περισσότερος χώρος ώστε ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη στη Συρία ως ανθρωπιστική κοινότητα βλέπουμε τις πιο τραγικές παραβιάσεις λόγω του πολέμου. 150 χρόνια μετά τη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού, στην επέτειό του αυτή, βλέπουμε το δίκαιο να καταπατιέται, να βομβαρδίζονται νοσοκομεία, να βομβαρδίζονται ε, νοσοκομιακά αυτοκίνητα, να ε, σταματούν τις εφοδιοπομπές του Ερυθρού Σταυρού, να σκοτώνουν τους οδηγούς. Βλέπουμε επίσης ορισμένους να λένε θα βοηθήσουμε αυτή την πλευρά με ανθρωπιστική βοήθεια και όχι, την, και το, όχι τους άλλους. Είμαστε υπέρ ημών και κατά των άλλων. Τόσο αντίθετο με το πνεύμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στις 18 Απριλίου εκδώσαμε ένα εντονότατο ανακοινωθέν τύπου το Συμβούλιο Ασφαλείας δηλαδή των Ενωμένων Εθνών που ανάγκασε το Συμβούλιο Ασφάλειας δηλαδή να πει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ακουστεί ως πολύ ισχυρή φωνή υπέρ του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα αυτό του ανθρωπιστικού χώρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε δράσεις για να ε, βοηθήσουμε τους σύρους. Θέλω να είμαι σαφέστατη. Ακόμα και αν οι ένοπλες σειράξεις σταματήσουν αύριο στη Συρία, οι πληγές είναι τόσο βαθιές που θα χρειαστεί η ανθρωπιστική βοήθεια εκεί για πολλά χρόνια. Και έρχομαι τώρα να πω το εξής. Ακούμε συχνά από ανθρωπιστικές οργανώσεις ένα απλό μήνυμα όταν ασκείται πίεση σε κάποια από τις δύο πλευρές, είτε στον Ασάντ είτε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να επιτρέψουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, ανταποκρίνονται. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε διαρκώς την έντονη αυτή πίεση. Το δεύτερο έχει σχέση με την παροχή πόρων, έτσι ώστε οι άνθρωποι εντός της Συρίας να λάβουν κάποια βοήθεια. Στην Ευρώπη διαθέσαμε 600 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς, Κομισιόν, 200 εκατομμύρια ευρώ και τα διαθέσαμε. Στην Ευρώπη ακόμα υπολοιπόμαστε ε, του να δώσουμε αυτά τα 600 εκατομμύρια και βεβαίως πρέπει να πράξουμε το καθήκον μας να προσφέρουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Επενώ το Κουβέιτ, το οποίο είπε θα διαθώσει 300 εκατομμύρια δολάρια και τα διέθεσε. Όμως από 1,5 δισεκατομμύριο υποσχέσεις τα μισά έχουν πραγματικά διατεθεί και γι' αυτό πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και διεθνώς να πράξουν οι δωρητές αυτά που υποσχέθηκαν. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας για να έχουμε στη διάθεσή μας τους πόρους που είναι απαραίτητοι. Σας λέω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και μέσα από τους παραδοσιακούς πόρους που διαθέτουμε, αλλά ταυτόχρονα να αναζητήσουμε και δημιουργικούς τρόπους να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους. Επίσης και λεπτομερίστερη περιγραφή των κυρώσεων κατά της Συρίας. Αλλά βεβαίως αυτά πρέπει να ωφελήσουν τον ίδιο τον Συριακό λαό. Εμείς θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το τρίτο και κρισιμότερο θέμα επί του παρόντος είναι η γειτονία. Εάν μέσα στην, στη Συρία υπάρχει πολιτική παράλυση, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος ωστόσο να μην κινητοποιηθούμε για να υποστηρίξουμε τις γειτονικέ χώρες έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος διασποράς. Και υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Φούλε και με τη δική μας ομάδα, επειδή αυτοί βλέπουν και τις ανάγκες αυτές πιο δραματικά, χαρτογραφούμε όλες τις δυνατές πηγές για να ε, αποσπάσουμε πόρους για να στηρίξουμε τις γειτονικές χώρες. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερα πράγματα. Χρειαζόμαστε ένα συνολικό στοχευμένο σύνολο μέτρων και τις δικές μας πηγές είτε και από άλλους δωρητές και οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί να κάνουν τι, να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες, νερό, ε, τρόφιμα, ε, στέγη, ιατρική περίθαλψη. Επίσης να στηρίξουμε τις κοινότητες των χωρών αυτών οι οποίες δέχονται πρόσφυγες και αυτό είναι κρίσιμο έτσι ώστε οι υπηρεσίες από την αποκομιδή των ε, σκουπιδιών μέχρι την παροχή νερού να φτάσουμε στους ανθρώπους αυτούς έτσι ώστε να αποφευθεί η διασπορά της βίας και επίσης και η μακροοικονομική σταθεροποίηση Είπατε πολύ σωστά, 3% είναι το κόστος. Εγώ βλέπω τα πράγματα αυτά στις χώρες αυτές με διαφορετικό μάτι, γιατί είναι πραγματικά δραματικές οι διαφορές. Όλοι συλλογικά μπορούμε να πράξουμε περισσότερα υπέρ των σύρων και υπέρ της περιοχής και πρέπει να κάνουμε περισσότερα, διότι πρόκειται για μια έκτακτη κρίση, μια εξαιρετική κρίση και η οποία απαιτεί έκτακτα μέτρα ως ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ, ευχαριστώ και εγώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Αυτή είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξη, με την ΤΕΒΕ. Η κυρία Ζολή. Ευχαριστώ την Επίτροπο, κυρία Γεωργίεβα, που ήρθε να μας μιλήσει, μας να, να μας μιλήσει για τις ε, εμπειρίες ε, της φρικτής κατάστασης στη Συρία και ιδίως στο Χαλέπι, όπου η, μεγάλη πλειοψηφία των γιατών έχει σκοτωθεί, απετέλεσε δηλαδή στόχο οι γιατροί, είναι μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση. Επίσης φοβόμαστε ότι ο Άσαντ έχει χρησιμοποιήσει χημικά όπλα κατά του πληθυσμού του και η έλλειψη ε, ε ψηφίσματος ε, από το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι δραματική. Υπάρχουν ε, χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι, εκτοπισμένοι από τα μέρη τους ε, και αυτό θα συνεχιστεί το φαινόμενο να αυξάνεται όσο υπάρχει ο Άσαντ πρόσφυγες που φεύγουν και ε, θέλουμε να δημιουργηθούν ακόμα ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Υπάρχει τεράστια πίεση στην Ιορδανία, στην Τουρκία και στο Λίβανο και όλη η περιοχή αντιμετωπίζει το κίνδυνο της αποσταθεροποίησης. Η παρουσία ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απολύτως αναγκαία και Είμαστε η πιο σημαντική ανθρωπιστική δύναμη στον κόσμο και κατά έναν τρόπο αντιστασμίζει αυτά όσα δηλαδή δεν κάνουμε από πολιτικής πτυχής. Πιστεύω ότι θα επιτύχουμε να όλοι μαζί να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν για να μπορέσετε να δράσετε. Όπως είπατε, τα τραύματα είναι τόσο βασιά που αυτά την πτώση του Ασάντ θα πρέπει να παραμείνουμε εκεί με την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι μία από τις πιο δραματικές καταστάσεις στον κόσμο σήμερα και την αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται μία ταυτόχρονη ανθρωπιστική καταστροφή και στη Σύρια και στο Μάλι και εφόσον γίνονται περικοπές στον προϋπολογισμό, ε, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε, να παράσχουμε τρόφιμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Γι' αυτό εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα πράτετε. Ο πρόεδρος κύριος Μπρόκ, ευχαριστώ κυρία Ζολή προτείνω να μιλήσουν όλοι δύο λεπτά μόνο, διότι πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς στις 5 και 40, διότι έχουμε το, την απονομή του βραβείου. Και το πρωτόκολλο είναι πανίσχυρο εδώ στο Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό δίνω το λόγο στην κυρία Γκόμες. Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για που μας παρουσιάσετε τόσο έντονα την κατάσταση. Και καταλαβαίνω το δίλημά σας και το δίλημά μας, ιδίως όταν αναφέρεται ότι κάθε ανθρωπιστικός νόμος παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, ε, ε, παραβιάζονται και από εμάς, τη Δύση. Εδώ πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξόντωσης και δεν νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία που, να συνεχιστούν αυτές οι φρικτές παραβιάσεις στη Συρία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς αξιολογείται την απόφαση που μόλις ελήφθη στο Συμβούλιο που ήρε τις κυρώσεις εκτός από το εμπάργο των όπλων. Ας πούμε ε, την εμπορία πετρελαίου στη Συρία. Και πώς αξιολογείται το, το ότι ετέθη ζήτημα παροχής όπλων από ορισμένα κράτη-μέλη και αν παρασχεθούν όπλα αυτό θα ε, χειροτερέψει ακόμα περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την πολύ λεπτομερή παρουσίαση. Καταλαβαίνω γιατί... But can I ask, if at some stage... Λέει ο κύριος Μπούτο Σιλ, μάλλον, και καταλαβαίνει γιατί χάνετε τον ύπνο σας. Μπορεί το κοινοβούλιο να συνεχίσει τον ύπνο του. Θα αφήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων στους ώμους κρατών που κάνουν διμερείς διαπραγματεύσεις. Τι θα γίνει με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, άμα θέλουμε να παράσχουμε πρέπει να υπάρχει και το περιβάλλον αποδοχής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπο, λέει κυρία Νίτς. Παρουσιάσατε με μαύρα χρώματα την εικόνα της Συρίας και το τι γίνεται εκεί και στις γειτονικέ χώρες. Πραγματικά φρίκι. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω από εσά είναι εάν αυτό το οποίο ζητάτε, μία συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για περαιτέρω στήριξη των γειτονικών χωρών, ε, συζητείται ή βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, στο Λίβανο που είχαμε πάει, όχι πρόσφατα σχετικά, η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει σε αυτούς τους οποίους προορίζεται τη λαμβάνουν. Παραδείγματος χάρη, ο, η, η η Μισέλινος βοηθάει στη Συρία ή έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ή γίνεται η παροχή της βοήθειας μόνο μέσω φορέων του ΟΗΕ. Επίσης, είναι πραγματικά απέσιο να παρακολουθούμε ε, τη χώρα μου, την Ολλανδία και άλλες χώρες όπου έγιναν δημόσιες ε, εκκλήσεις χρηματοδότησης ε, να βλέπουμε μια τόσο πενιχρή ανταπόκριση του πληθυσμού στις εκκλήσεις χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι πολύ λυπηρό και αυξάνει την ευθύνη που έχουμε εμείς τους ώμους μας. Κυρία Σαργεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν επισκεφθήκε την Ιορδανία η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στα σύνορα με τη Σύρια του Φεβρουάριο, ένας εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας είπε, με εξέπληξε αλλά το μην μιλάτε για επανεγκατάσταση εκτός σε χώρες εκτός περιοχών της. Μην μιλάτε για επανεγκατάσταση στην Ευρώπη, γιατί θα αυξήσει τον αριθμό όσων φεύγουν από τη Συρία και που βρίσκονταν τότε στην Ιορδανία. Αυτό ήταν μια κοινική παρατήρηση, αλλά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της επανεγκατάστασης ιδίω μετά την πτώση του Ασάντ θα φύγουν από τη Συρία πρόσφυγες που δεν θα γυρίσουν πίσω, δεν θα γίνονται δεκτοί στη χώρα αυτή, ούτε θα γίνονται δεκτοί στις γειτονικέ χώρες. Έχετε ιδέες για το τι θα γίνει. Ξέρω ότι είναι αρμοδιότητα της κυρίας Μάλστρομ, αλλά θα πρέπει να δούμε το θέμα της επανεγκατάστασης των Σύρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερη ερώτηση. Κατά την άποψή σας υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ασφαλών ζωνών στη Συρία. Γίνεται μια σχετική συζήτηση. Λένε άλλοι ότι είναι κακό γιατί εκεί βρίσκεις περισσότερα πιθανά θύματα. Τι λέτε εσείς. Τρίτον, Παλαιστίνοι πρόσφυγες που φεύγουν από τη Συρία, φεύγουν για δεύτερη φορά στη ζωή τους ενδεχόμενα, δηλαδή η οικογένειά τους ε, είχε φύγει είτε το 48 είτε το 67 και αποτελούν βάρος και στην Ιορδανία που δεν τους αφήνει να μπουν και στο Λίβανο. Υπάρχει ένας φόβος ότι θα αποσταθεροποιήσουν τις χώρες αυτές. Τι κάνετε με το Παλαιστινιακό, με το θέμα δηλαδή, των Παλαιστινίων προσφύγων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ομάδα μου με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ θέλει να ζητήσει την κατάπαυση του πυρός των ε, πλευρών ζητών, αναζητώντας μια, μια θέση με διαπραγμάτευση. Εμείς είμαστε υπέρ των πολυμερών ε, συζητήσεων για να δοθεί απάντηση στις, ε, στα ζητήματα στη Συρία και να ξεκινήσει μια συντακτική διαδικασία στην οποία θα εμπλέκεται και ο πληθυσμός αυτός. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφευθεί η ανθρωπιστική καταστροφή. Μας ανησυχούν οι πληροφορίες της 27ης Μαρτίου όταν ε, στο, σε ένα στρατόπεδο στην Τουρκία, της στην Σουλεϊμάνδια, έγινε διαδήλωση κατά των συνθήκων ζωής των ε, προσφύγων και μετά από την ε, διαμαρτυρία αυτή 427 άτομα ξαναστάλθηκαν πίσω στη Συρία κατά παραβίαση των αρχών της μη επαναπροώθησης. Επίσης μας ανησυχεί η συγκεκριμένη περίπτωση των Παλαιστινίων στη Συρία διότι γίνονται στην πραγματικότητα διπλά πρόσφυγες και θα πρέπει να έχουν ειδική αντιμετώπιση και μία παρακολούθηση από πλευρά της διεθνού κοινότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Δύο βασικές ερωτήσεις για την κατάσταση των προσφύγων. Πρώτον, χριστιανοί, ιδίως μετά την ε, φρικτή απαγωγή των επισκόπων. Και δεύτερον, και όπως είπε και κάποιος πράσινο συνάδελφος. Πολλοί από αυτούς είναι διπλά πρόσφυγες. Οι χριστιανικές κοινότητες δεν είναι μόνο παλιοί, αλλά και κάποιοι που έφτασαν ως πρόσφυγες από το Ιράκ. Δεκάδες χιλιάδες χριστιανοί του Ιράκ είναι πρόσφυγες στη Συρία και τώρα βρίσκονται σε διπλό κίνδυνο. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για περιπτώσεις που υπάρξει που κυριαρχήσουν οι εξτρεμιστές. Επίσης, Hezbollah. Η ομάδα μου θεωρεί ότι το Χεσμολά είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες ότι το Χεσμολά, οι μονάδες του, εμπόδισαν πρόσφυγες να περάσουν στο Λίβανο ή έστειλαν πίσω πρόσφυγες στο, από το Λίβανο. Έχετε πληροφορίες. Ήταν πρόσφυγες εν γέννη, ήταν χριστιανοί μόνο. Και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτή τη φρικτή συμπεριφορά του Χεσμπολά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στο Μάλι πολεμούμε τους ε, τρομοκράτες και τις τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες ε, έχουν ένα στοιχείο φαμενταμελισμού. Ε, τι κάνουμε στη Συρία. Έχουμε εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε ο εξοπλισμός με τον οποίο υποβοηθούμε τις εντατικές ομάδες δεν θα περιέλθει σε ακραίες ομάδες. Δεύτερο θέμα. Απήχθησαν σήμερα δύο Μητροπολίτες ε, Ελληνοορθόδοξος και Συροορθόδοξος. Ε, θα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργήσουμε εις τρόπον ώστε να υποβοηθήσουμε την απελευθερωσή της. Και τρίτον, το γενικότερο θέμα της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή η οποία έχει ε, και έχει λάβει ε, χαρακτήρα ε, γενικής επίθεσης κατά των χριστιανών. Ε, προτιθέμεθα να διατηρήσουμε τις κάποιες ισορροπίες σε σχέση με τους χριστιανούς στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, uh, Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ λέει κυρία Κοπά. Ε, μας μιλήσατε για ένα πραγματικά μια ανθρωπιστική τραγωδία ε, ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά ε, στις, στις χρηματικές, στις πιστώσεις. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα όσον αφορά τη διάθεση επαρκών πιστώσεων. Έχετε ταυτοποιήσει νέους δωρητές, νέους νέες πηγές χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πολλά ακούμε, λίγα γίνονται έχουν ανταποκριθεί όλοι οι προσφέροντες, ας πούμε άτομα, ιδιώτες, οι φορείς, ιδρύματα κλπ. Και πιστεύω επίσης ότι μέτρα πρέπει να ληφθούν και στο Λίβανο και στην Ιορδανία για να μην δημιουργηθούν ε, ρατσιστικές συγκρούσεις, ένα περιβάλλον ρατσιστικό κατά των προσφύγων. Συμφωνώ πάντως απολύτως με σας αυτό που έχει απόλυτη προτεραιότητα είναι η υλοποίηση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, διότι αυτό που βλέπουμε τώρα στη Συρία μας γυρίζει πίσω δεκαετίες πολλές. Ο, ο πρόεδρος, ο κύριος Ρότα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κατάσταση δεν μπορεί να Κυρία Επιτροπή, η κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει. Μιλάμε όλοι για ανθρωπιστική καταστροφή. Μιλήσατε για ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Πώς θα εξασφαλίσετε την ασφάλεια αυτών των περιοχών. Άλλες χώρες, η Ορδανία για παράδειγμα, που έχει κοντά 400.000 ε, πρόσφυγες και ακούγεται ότι θα τριπλασιαστεί μέχρι το τέλος του έτους ο ρυθμός των προσφύγων εκεί. Μέχρι πού θα φτάσει. Μιλάμε για μια ανθρωπιστική κατάσταση. Πεθαίνουν άντρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο με χρήματα και θα, που θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση γιατί το πρόβλημα θα περάσει σε μια άλλη χώρα, θα ξαναγίνουν ανθρωπιστικές προσπάθειες, αλλά χρειάζεται μια πιο ισχυρή μορφή παρέμβασής μας. Η κυρία Γκρέις, ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι για την ανθρωπιστική προσπάθεια της Ένωσης στη Συρία και θέλω να επενέσω εκ νέου το έργο της κυρίας Γεωργίευα στον τομέα, αλλά δεν πιστεύω ούτε στιγμή ότι η λύση της κρίσης στην Συρία θα λυθεί αποκλειστικά σε ανθρωπιστικό επίπεδο, αλλά που χαρακτήρα. Δείξατε, υπογραμμίσατε την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και στις χώρες γύρω από τη Συρία, ιδίως ε, λόγω των διωγμένων πληθυσμών. Ξέρουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ε, οι γυναίκες πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα. Η ερώτησή μου είναι υπάρχουν ειδικέ δράσεις και ανέπιες ναι, για γυναίκες. Ευχαριστώ. You're forgiven this time. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας καλωσορίζω κύριε Επίτροπε και σας ευχαριστώ πολύ για τις δεσμεύσεις σας ε, και τα ειλικρινά σας λόγια και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ σημαίνει για αυτή την κατάσταση ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη στο Λίβανο και ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως η χώρα αυτή έχει απορροφήσει ένα εκατομμύριο σχεδόν πρόσφυγες. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο αυτό θα υποστηρίξει την παροχή όλων των μέσων που χρειάζονται και θα πιέσει και την ε, ψήφιση, την ε, υιοθέτηση ενός ψηφίσματος τον ερχόμενο μήνα. Πρέπει να τονίσουμε την παρουσία λίγων αλλά πολύ επικίνδυνων τζιχαδιστών, ακραίων ε, Ισλαμιστών δηλαδή, στην Συρία. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ακραίους ε, και τους φονταμεταλιστές ε, με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι χρήματα χρειάζονται για την βοήθεια αυτή. Θα ήθελα να ξέρω πόσα χρήματα θα δαπανηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα δαπανηθούν και έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη στις παροχές. Επίσης, πώς θα ενθαρρύνουμε ε, τις χώρες του ραβικού τις αραβικές χώρες και του αραβικού κόλπου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια επίπτωση μετά από εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά την πρόσβαση στους ε, θυγόμενους και σε αυτούς που έχουν ανάγκη ε, παροχής βοήθειας. Και τέλος πρέπει να, να ζητήσουμε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ για να αποφευχθεί η εξάπλωση του προβλήματος στο, Λίβατο, στο Λίβανο. Βεβαίως πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, κοινότητες, ε, αλλά δεν είναι το ίδιο όσο η αποστολή μιας ειρηνευτικής δύναμης για ειρήνη και σταθερότητα. Δεν είναι το ίδιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Επίτροπος. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτήν την πολύ, αυτή τη συζήτηση που γίνεται σε βάθος και με ειλικρίνεια και θα ήθελα να απαντήσω καταρχάς στην κυρία Ζολή. Αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονες τραγωδίες και στην ανθρωπιστική κοινότητα και στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε αυτό το φοβερό δίλημα θα βοηθήσουμε όλο και περισσότερο τη Συρία εις βάρος άλλων που έχουν ανάγκη ε, ε, δέχτηκα τον ε, μεταβατικό ηγέτη της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας η οποία και αυτή βρίσκεται σε μια φρικτή κατάσταση και χρειάζεται άμεση βοήθεια την προσωρινή ηγεσία. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να, να τραβήξουμε, να τεντώσουμε ε, τις δυνατότητες που έχουμε, τα μέσα που έχουμε ε, για να τα διαθέσουμε σε, σε όλες αυτές τις ε, καταστάσεις αλλά με τον καλύτερο τρόπο. Η κυρία Γκόμες έθεσε δύο πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Η οι συγκεκριμένες κυρώσεις ε, θα βοηθήσουν. Αυτό εξαρτάται. Αποφασίστηκε ότι με αυτόν τον τρόπο της άρσης δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την αντιπολίτευση, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε τους, τον πληθυσμό που βρίσκεται σε μέρη τα οποία ελέγχει η αντιπολίτευση. Γι' αυτό που ζήτησαν να συζητήσουμε ακριβώς το θέμα αυτό ε, στην επιτοπή που είναι αρμόδια για τις κυρώσεις. Αν απελευθερωθούν πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι διοχετεύονται ε, σίγουρα 100% στους δικαιούχους. Το δικό μου αίτημα ήταν να προσφέρουμε τα μέσα τα δικά μας, τη γνώση μας όσο μπορούμε καλύτερα. Βεβαίω χρειαζόμαστε περισσότερα πιστώσει, περισσότερα κονδύλια για μια κατάσταση η οποία επιδεινώνεται δραματικά. Δεν υπάρχουν λιπάσματα. Χωρίς λιπάσματα δεν υπάρχουν σοδιές. Δεν υπάρχουν χημικά για, να, ε, για, το, για το πόσιμο νερό, για να καθαρίσουν το νερό ώστε να είναι πόσιμο δεν υπάρχουν ε, τα, τα αναγκαία μέσα για, την παραγωγή προϊόντων. Λοιπόν, ε, ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και σας ευχαριστώ για την δική σας παρέμβαση. Για τα, έπλα, για τα όπλα. Εγώ μιλάω για την κατάσταση μέχρι σήμερα. Μπορεί να αλλάξει αύριο. Για τα όπλα. Η μόνη χρήση όπλων που έχει χρησιμοποιηθεί ως ανασχετικός παράγοντας ήταν η πύραυλη Patriot στην Τουρκία. Ανασχετικός παράγον. Ε, μέχρι τώρα περισσότερα όπλα δεν έχουν οδηγήσει στο να συνετιστούν οι αντικρυόμενες πλευρές και να κάτσουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Δεν έχει οδηγήσει σε αυτό καθόλου, αλλά δημιούργησε περισσότερες και περισσότερη βία. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι αυτή η εξίσωση πρέπει να αλλάξει και έτσι θα υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλά εμείς ως ανθρωπιστές ανησυχούμε επειδή δεν βλέπουμε επαρκή ενέργεια να διατίθεται, επαρκή προσπάθειες να γίνονται για τη διαπραγμάτευση. Πολλοί είπαν ότι μόνο μέσω πολιτικής οδού μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της τραγωδίας της Συρίας. Όσοι το είπαν αυτό έχουν δίκαιο. Αυτό είναι σωστό. Μπορούμε να πούμε, όσο και δύσκολη να είναι μία τέτοια λύση, πρέπει να την υποστηρίξουμε και χτες στο Συμβούλιο Εξωτερικών, Υπουργών Εξωτερικών, πολλά κράτη-μέλη επέμειναν και είπαν ότι υποστηρίζουν την πολιτική λύση. Ο κύριος ε, Μίτσελ ε, ρώτησε εάν μπορούν να δημιουργηθούν ε, ασφαλείς ζώνες όπου μπορεί να παρισχεθεί και να διατεθεί ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστική διάδρομη. Στο, στην παραμεθόρια περιοχή με την Τουρκία υπάρχουν άνθρωποι που ε, επιβιώνουν σε, μια, σε μια κατάσταση η οποία έχει λιγότερη βία από ό,τι είχε, αλλά δεν είναι βεβαίως καλή αυτή η λύση. Υπάρχουν διάφορες ζώνες όπου παρατηρείται λιγότερη βία. Η εμπειρία μας από το παρελθόν δείχνει ότι αυτή η δημιουργία ζωνών δεν είναι καλή λύση. Γιατί, διότι χρειάζεστε κάποιον να προστατεύσει, να ε, ε, εποπτεύει αυτές τις ζώνες όπως ε, λέμε μπότε στο έδαφος, δηλαδή κάποια δύναμη την οποία δεν έχουμε. Και πολλές φορές αυτές οι δίθεν ασφαλείς ζώνες ε, γίνονται heavens, buffer zones being actually turned into... θύλακες, θύλακες ε, ομοιρίας και πολλές φορές χρησιμοποιούνται από μαχητές για να έρθουν να ξεκουραστούν για λίγο, για να ξαναρχίσουν τη μάχη. Δεν έχουμε δυστυχώς ε, ειρηνευτικές δυνάμεις, ούτε ειρηνευτικό δυναμικό αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε, ε, δεν πιστεύουμε, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή πεπισμένοι ότι υπάρχει νευτική λύση για τη Συρία. Όχι ότι εγώ θα αρνηθώ οποιαδήποτε πρόταση, αλλά πρέπει να ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες. Αν προτείνεται νευτική δύναμη, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς υπό ποιες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή δεν διαβλέπουμε μια τέτοια λύση. Όσον αφορά τώρα τις ε, ασφαλείς ε, οδούς ε, του ασφαλεί διαδρόμου παροχή. Ένα διάδρομο από πού προ πού. Πώ προστατεύουμε αυτή την οδό, αυτό το δρόμο. Ούτε αυτό είναι μια λύση που μπορούμε να εξετάσουμε. Αυτό που την παρατήρηση της κυρίας Νέιτς. Εάν η ανθρωπιστική βοήθεια ε, φτάνει στους αποδέκτες όλους. Όχι με τις καλύτερες συνθήκες από 6,5 εκατομμύρια που χρειάζονται μπορούμε εμείς να τη δώσουμε σε 2 εκατομμύρια με τις καλύτερες συνθήκες και εκεί όπου μπορούμε σήμερα να δώσουμε βοήθεια μπορεί αύριο να μην μπορούμε να πλησιάσουμε αυτό που αναγνωρίζουμε είναι ότι εδώ δεν συζητάμε μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πέραν αυτού και υπεράνω αυτού μιλάμε για το 2% που ανέφερε ο κύριος Μπροκ. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν και οι γειτονικέ χώρες και να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετες πιστώσεις Ποιο έχει τώρα, πώ κρατάει στα χέρια του τι πρόσθετε πιστώσει και πώς μπορούμε να του πιέσουμε. Εκεί υπάρχει προσπάθεια να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και πραγματικά με τους συναδέλφους πηγαίνω παντού. Χτες στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και τους δείχνω αυτό το πίνακα και εσείς τον πήρατε. Είναι το ε, επικαιροποιημένο brief για τη Συρία. Στην τελευταία σελίδα λέει, βλέπετε ποιος δεσμεύτηκε να δώσει τι και πόσα. Θετικό είναι το ότι προσθέτουμε πράγματα. Χτες ανέφερα τις πέντε χώρες που έδωσαν περισσότερο από 10 εκατομμύριο ευρώ. Και αμέσως δύο υπουργοί είπαν και εμείς είμαστε εκεί, και εμείς είμαστε εκεί. Το ίδιο κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε με άλλους. Κυρίως κοιτάμε, όποιος είπε θα δώσω 300 εκατομμύρια, να δώσει 300 εκατομμύρια. Η Ρωσία δεν, έδωσε, δεν δεσμεύτηκε τίποτα. Η Κίνα μόνο για κάτι συμβολικό σχεδόν. Ζητώ από τα Ηνωμένα Έθνη να είναι πιο δραστήριοι στο name and shame, στον κατομονόμασμό των χωρών, διότι η κρίση είναι παγκόσμια. Μετά, το θέμα είναι και το τι κάνουμε με τα χρήματα αυτά. Βάζουμε 200 εκατομμύρια από την Επιτροπή. Τι αντίκτυπο έχει. Βοηθούμε αυτούς που παρέχουν τροφή υγειονομική περίθαλψη, προστασία και αυτό για πολλούς είναι σωτήριο. 50, έτσι όπως το έχουμε κανονίσει είναι 50% των ε, πόρων πηγαίνει για τη Συρία, στο εσωτερικό της Συρίας, το 50% εκτός. Το, η Πατερμοστία, το, παγκόσμιο, το παγκόσμιο πρόγραμμα επιστημισμού έχουν συμβάλει το 50% μέσα στη Συρία είμαστε αποφασισμένοι να το μοιράσουμε 50-50 σε κυβερνητικές περιοχές, σε περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες. Κοιτάζουμε κάθε οδό μεταξύ των οποίων να, αν μπορούμε να περάσουμε βοήθεια μέσω των τουρκικών συνόρων, το κάνουμε. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι ό,τι και να κάνουμε συνεχίζει να παραμένει η απόκληση. Και επανέρχομαι σε αυτό που πολύ είπατε. Η λύση είναι πολιτική. Είναι άδικο προς τους ανθρώπους που παρέχουν την ανθρωπιστική βοήθεια να, και που διακινδυνεύουν πολύ τη ζωή τους να τους λέμε κάντε τη δουλειά σας, δεν είναι δική μας δουλειά να σας ε, προσφέρουμε υποστήριξη. Για το θέμα της επανεγκατάστασης. Κύριε Σαργεντίνη, τα κράτη-μέλη της Ένωσης σε, ατομικό, σε ατομική βάση και σε θελούσια βάση δεσμεύτηκαν για 50.000 άτομα με προσωρινή προστασία, σύρους. Εγώ γνωρίζω ότι είχαμε περιπτώσεις όταν μια πρώιμη, μια πρόορη αποδοχή της επανακατάστασης οδήγησε σε αύξηση, αύξηση των προσφύγων. Στην Ταϊλάνδη, για παράδειγμα. Στην περίπτωση εκείνη, όσοι έφυγαν για επανεκατάσταση μείνανε. Λέμε λοιπόν και στο UNHCR ότι δεν θέλουμε να υπάρξει ένας παράγοντας έλξης που να οδηγεί στα κράτη στο να είναι πιο ε, να καθυστερούν περισσότερο. Ξέρω ότι πρέπει να τελειώσω. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα πιο συλλογικά, συμφωνώ. Παλαιστίνη. Ήταν 500.000 στη Συρία, εκ των οποίων οι 400.000 ε, θέλουν βοήθεια. 45.000 έχουν φύγει. Στο Λίβανο κυρίως, σε άθλιες συνθήκες κατά βάση χριστιανοί. Όλες οι μειονότητες, όχι μόνο χριστιανικές μειονότητες, αισθάνονται ότι απειλούνται. Και η απαγωγή των επισκόπων είναι ένα φρικτό γεγονός όντως. Συνεργαζόμαστε με εταιρούς ούτως ώστε να δοθεί προσοχή στις πιο επικίνδυνες κατηγορίες. Ηλικιωμένοι, γυναίκες, παιδιά και μειονότητες βέβαια. μπορώ να σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιγόντως κάθε κατηγορία που βρίσκεται σε κίνδυνο. Και θα ξανάρθω αν θέλετε γιατί βλέπω ότι δεν, έχετε, δεν έχουμε χρόνο. Η Αυστρία έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια διαθρησκιακού διαλόγου στη Συρία και νομίζω ότι θα έπρεπε να υποστήριξουμε περισσότερο όντως αυτούς που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Γυναίκες. Ήμασταν πρωτοπόροι στο να κάνουμε το gender marking της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην Συρία βλέπουμε μαζικοποίηση του βιασμού και εντάξαμε μαζί με την ύπατη τη διάσταση αυτή στο πλαίσιο της προστασίας ιδίως λόγω και της μαζικής ε, παρουσίας προσφύγων. Τώρα η εντολή του ΟΗΕ το ψήφισμα του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια νομίζω τώρα είναι πιο αποτελεσματικό από ό,τι ήταν πριν από λίγους μήνες γιατί όλοι καταλαβαίνουν το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά αν δεν υπάρξει πίεση από πλευρά μα θα χαθεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος και τελειώνω. Πόσοι Ευρωπαίοι πέθαναν για να υπάρξει ε, οι διεθνείς, ε, να υπάρξουν διεθνείς συμβάσεις για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση του πολέμου. Ο πρόεδρος Μπροκ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Βλέπετε και οι ακούτε από τα χειροκροτήματα που δεν έχουν πάντα την τύχη να ακούν μετά τις δηλώσεις τους οι επίτροποι ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών βλέπετε την υποστήριξη. Και γι' αυτό ενθαρρύνομαι να σας προτείνω να προσπαθήσω μαζί με την κυρία Ζολή της Επιτροπής Αναπτύξεως και του κυρίου Λαμασούρ των προϋπολογισμών να συντάξουμε κοινή επιστολή που να απευθύνουμε στο Συμβούλιο Υπουργών και στην Κομισιόν για να ζητήσουμε ενίσχυση της χρηματοδοτικής υποστήριξης των προσφύγων στην Σύρια. Αν συμφωνείτε θα αναλάβω αυτή την πρωτοβουλία. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτροπή.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 Ladies and gentlemen, may we invite you to sit down. President Schulz is... Σας παρακαλούμε, παρακαλώ, ε, παρακαλώ να καθίσετε. Έρχεται ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς. gentlemen, please take your seat. Ο πρόεδρος Μπροκ, καθίστε σας παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσει το θέαμα εντός ολίγου. Επιλέξει. Use the hammer. Throwing. So, but they are in front of the door now. They are coming now with President Schultz. Is the music playing? Die internationale? Frau Schulz. But we have not done the Ο πρόεδρος Μπροκ. Κυρίες και κύριοι, ορίσατε και παρακαλώ απευθύνετε μαζί μου χαιρετισμό και ορίσατε στις βραβευθύσεις του 2005 το βραβείο Ζαχάροφ της κυρίας με τα Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που διεξάγουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Αναπτύξεως και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτ τον οποίον <clears throat> υποδέχομαι εδώ και απευθύνω χαιρετισμό. Πέρασε καιρός μέχρι ότου έχουμε την ευκαιρία απονομής του βραβείου και ελπίζω ότι αυτό ωστόσο θα εκλειφθεί ως καθαρό μήνυμα τη συμπαράστασή μα σε όσου αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο απανταχού του κόσμου και για το θάρρο που δείξατε απέναντι που διοικεί τη χώρα σα. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκεστε σήμερα εδώ κοντά μας θα δούμε ένα μικρό, μια μικρή ταινία για την απονομή του βραβείου τότε, το 2005, όπου δυστυχώς ήσασταν απούσες. Siguen caminando. Otra vez hemos venido y queremos entregar aquí, que es una manera personal, no atención a la población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 no se encuentran hoy, desgraciadamente, con nosotros. Nosotras no recogeremos el premio hoy. Das Wort hat der Präsident des Europäischen Παραδίδω το λόγο στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Είναι μεγάλη η χαρά που με διακατέχει που υποδέχομαι σήμερα τις κυρίες λευκά στις οποίες απονομήθηκε το βραβείο Ζαχάροφ το 2005. Νομίζω στο όνομα όλων σας αλλά και στο όνομα όσων δεν είναι σήμερα εδώ τις καλωσορίζω. Για μας είναι ιδιαίτερη η ημέρα η σημερινή που βρίσκεστε εδώ κοντά μας σήμερα και συμμεριζόμαστε τη συγκίνησή σας. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για τους ευρωβουλευτές. Το βραβείο Ζαχάροφ 2005 είχε απονομηθεί το ίδιο έτος και στον Ανουάρ Ιμπραήμ και στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, των οποίων εκπρόσωποι παρελίστανται σήμερα. Και το βρίσκω πολύ όμορφο αυτό, ότι βρίσκονται δηλαδή σήμερα εδώ και οι άλλοι βραβευθέντες του έτους 2005 και απευθύνω και σε αυτούς θερμό καλώς ορίσατε. Για λόγους εκτός δικού μας αλλά και δικού σας ελέγχου η απονομή του βραβείου του 2005 δεν μπόρεσε να γίνει με δική σας παρουσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν βραβεύει την διαρκή ειρηνική μάχη, τον διαρκή ειρηνικό αγώνα των κυριών με τα λευκά στην Κούβα. Εκτιμούμε την δέσμευσή σας για την προστασία των δικαιωμάτων και έχετε επιλέξει το λευκό χρώμα που συμβολίζει την ειρήνη. Με την άρνηση των κουβανικών αρχών να σας επιτρέψουν την μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραλάβετε το βραβείο, ήδη και γι' αυτό, ήδη και με αυτό παραβιάστηκε θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμά σας. Αυτό δηλαδή που περιλαμβάνεται ως αρχή στην διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ότι κανείς μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να εγκαταλείψει τη χώρα του και να επανέλθει σε αυτήν. Ως θαραλέες και επίμονες γυναίκες, και γι' αυτό απευθύνομαι ειδικά σε εσά της τέσσερις κυρίες εδώ μπροστά μου και εσάς εδώ δίπλα μου. Ως λοιπόν θαραλέες και επίμονες γυναίκες έχετε συνηθίσει ωστόσο να διανύετε μακρές αποστάσεις. Ο δρόμος από την Κούβα έως τις Βρυξέλλες κράτησε παραπάνω από 7 χρόνια. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να σας απευθύνω το καλό ορίσατε, γιατί αυτά τα 7 χρόνια δείχνουν ότι καμιά δικτατορία στον κόσμο δεν μπορεί να αποτρέψει την δημοκρατία στο διηνεκές. Γι' αυτό χαίρομαι τόσο πολύ που είστε σήμερα κοντά μας. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι αυτό για σας και Αυτά που θα πω τώρα θα είναι και τα πιο δύσκολα για σας. Η συνειδρήτρια και τότε επικεφαλής της ομάδας σας, των κυριών με τα λευκά, η Λάουρα Ινές Πολέδο απεβίωσε το 2007. Δεν μπόρεσε δηλαδή να έλθει μαζί σας στον δρόμο αυτό. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό που ναι μεν η Λάουρα ίδια δεν είναι σήμερα εδώ, το πνεύμα της όμως σίγουρα βρίσκεται εδώ. Δεν την έχει λησμονήσει κανείς. Προ δεκαετίας, όταν, αγαπητή Βέρτα, ο σύζυγός σας, όταν προ λοιπόν, αγαπητή Βέρτα, ο σύζυγός σας, αλλά και της Λάουρα, ο σύζυγος Γκουτιέρες, συνελήφθησαν στη διάρκεια της Μαύρης Άνοιξης, αποφασίσατε εσείς οι δύο να αντιδράσετε ειρηνικά κατά της αυθαίρετης αυτής της σύλληψης. Αυθόρμητα προσήλθαν πολλές σύζυγοι, μητέρες και θυγατέρες ακτιβιστών και διαμαρτυρηθήκατε καθημερινά στους δρόμους της Σαββάνας απαιτώντα την απόλυση όλων των πολιτικών κρατουμένων, πράγμα το οποίο κάνετε μέχρι σήμερα. Από τότε λοιπόν ο ελληνικό σας αγώνας κυριαρχεί ως σύμβολο της κουβανικής αντίστασης κατά της κουβανικής κυβέρνησης, μιας κουβανικής αντίστασης υπέρ της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Χιλιάδες γνωστές και άγνωστες κουβανές υποστηρίζουν την προσπάθειά σας. Θα ήθελα τώρα να αποτίσω φόρο τιμή σε δύο, ο Σβάλτο Παγιά και Φαρίνας, που ήταν οι βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχαρόφ του 2002 και 2010. Ο Σβάλτο Παγιά σκοτώθηκε πέρσι σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ωστόσο, οι ιδέες του ζουν και θα συνεχίζουν να ζουν. Και ο ίδιος και η μνήμη του θα εμπνέουν μελλοντικέ γενναίες κουβανών ακτιβιστών και ακτιβιστριών και θα σας ενθαρρύνουν να μην παρατήσετε τον αγώνα. Αγαπητές συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνουμε ότι ο Ραούλ Κάστρο έχει αναλάβει πολλές μεταρρυθμίσεις φιλελευθερωποίηση της οικονομίας, ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, άνοιγμα της αγοράς. Αλλά παρά τις μεταρρυθμίσεις αυτές και παρά ή ίσως και ελπίζω στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων αυτών που υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις ωστόσο η Κούβα είναι η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που αρνείται οποιαδήποτε μορφή πολιτικής αντιπολίτευσης. Κάποιες μεταρρυθμίσεις μπορεί να έγιναν, δεν συμβαδίζουν όμως με πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Θα σας θυμίσω τα εξή νούμερα. 2012 η Κουβανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικής Συμφιλίωσης σημειώνει συνολικά 6.602 περιπτώσεις αυθαίρετης σύλληψης μικρής χρονικής διάρκειας. 50% περισσότερες από το 2011. Το 2013 ακολουθεί μέχρι τώρα πάνω από 1.200 συλλήψεις. Η δική μου προσωπική άποψη, αλλά νομίζω ότι απηχώ και την άποψη των περισσότερων ευρωβουλευτών, είναι σαφής. Εάν η κουβανική ηγεσία θεωρεί ότι είναι αρκετά ισχυρή και έχει την άποψη ότι νομιμοποιείται πολιτικά να δράμε τον τρόπο αυτό. Εάν θεωρεί ότι διαθέτει την πλήρη υποστήριξη του λαού, εάν όντως πιστεύει αυτά τα οποία δηλώνει προς τα έξω, ότι ολόκληρη Κούβα την υποστηρίζει, τότε πραγματικά δεν χρειάζεται τέτοια νούμερα. Δεν χρειάζεται καμιά αυθαίρετη σύλληψη, δεν χρειάζεται καμιά καταπίεση της αντιπολίτευσης. Εφόσον κάποιος αποφασίζει να υλοποιήσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, αυτό σημαίνει ότι αισθάνεται αρκετά ισχυρός, ότι δεν φοβάται τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, ότι δεν έχει τον λαό αντίθετό του. Όποιος καταπιέζει τον λαό, αυτός φοβάται τέτοια πράγματα. Όποιος όμως φοβάται τον λαό, έχει και λόγους να τον φοβάται. Και ποτέ δεν θα μπορέσει να κερδίσει, διότι κανείς λαός δεν δέχεται επάπειρον την καταπίεση το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, το δικαίωμα της ελευθερίας σκέψης, το δικαίωμα της ελευθερίας κίνησης είναι θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να εμποδίσει τους πολίτες αυτούς να αγωνιστούν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών. Εν τέλει δε να νικήσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί σχέσεις με την Κουβανική Εθνοσυνέλευση μέσω της Ευρωλάτ αλλά και μέσω του Παλατίνο, του Παρλατίνο του Λατινοαμερικανικού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε διαρκή και δραστήριο διάλογο με την αντιπολίτευση. Και η στήριξη προς αυτή την αντιπολίτευση για μας συμβολικά είναι δυνατόν αυτό με την απότηση φόρου τιμής σε εσά σε εσά που βρήκατε τρόπους να εκφράσετε την άποψή σας υπό δυσχερή συνθήκες. Αναμένουμε μαζί σας την ημέρα όπου και άλλοι κουβανοί και άλλες κουβανές θα μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς φόβο αντιπίνων. Ελπίζω και εύχομαι η ημέρα αυτή να εξασφαλιστεί σύντομα για όλους τους κουβανούς και όλες τις κουβανές. Πιστεύω απόλυτα ότι η ημέρα αυτή θα έλθει. αγαπητές κυρίες με τα λευκά, στον δρόμο προς την ελευθερία, στον δρόμο προς τη δημοκρατία, έχετε καλύψει μεγάλο διάστημα. Σήμερα περνάτε από τις Βρυξέλλες. Να είστε βέβαιες ότι βαδίζουμε μαζί σας. Και με μεγάλη μου χαρά, με καθυστέρηση μεν, αλλά σήμερα πραγματικά, σας απονέμω σήμερα το βραβείο Ζαχάροφ του 2005.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 Un Ευχαριστώ και χαιρετώ τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τους παρόντες βουλευτές. Καταρχάς δεν έχω λόγια. Θα ήθελα να ζητήσω να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή σε ανάμνηση της Λάουρα Πογιαντολέδο που ήταν βραβείο Ζαχάροφ αλλά και για τον Εδάδο Παγιάν Χαρδίνιο που ήταν αγωνιστές της δημοκρατίας που έχασαν τη ζωή τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Παρακαλώ ένα λεπτό σιγής για όλους αυτούς. Σε, Κυρίες και κύριοι, είμαι εδώ εξ ονόματος των ε, κυριών με τα λευκά. Θέλω καταρχάς να σας πω ότι θα ήθελα το βραβείο αυτό να το δεχθεί η Λάουρα Πογιάν, γυναίκα που δεν είναι εδώ μαζί μας. Μια γυναίκα που ήταν η εμπνεύστρια του κινήματός μας, μια κυρία. Αυτά που λέω εγώ όμως τώρα εδώ εξ ονόματος ε, των γυναικών εικόν ε, με τα λευκά θα τα διαβάσει η κόρη της, η Μαρία Λάουρα Πογιάν. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι μεγάλη τιμή για μας να έρθουμε ενώπιόν σας για να δεχθούμε αυτό το βραβείο που εμπνέεται από την μνήμη του Αντρέη Ζαχάροφ που ήταν έμπνευση για την ειρηνική μάχη μας. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι παίρνουμε το βραβείο αυτό στο όνομα όλων των γυναικών που μετέχουν στο, στο κίνημά μας, χωρίς την θυσία των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η δική μας παρουσία εδώ. Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, ουδέποτε ωστόσο χάσαμε την πίστη στο ότι κάποια μέρα θα ήμασταν εδώ για να σε ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας και για να εξηγήσουμε την νίκη μας. Είμαστε μητέρες, σύζυγοι, παιδιά, μέλη των οικογενειών κουβανών που είναι στην φυλακή γιατί διεκδικούν το βασικό δικαίωμα ενός ανθρώπου, να ζήσουν με βάση τη συνείδησή τους. Είμαστε πάνω απ' όλα γυναίκες που δραστηριοποιούμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, που αγωνιζόμαστε στη μάχη για, για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας, καλύτερο από αυτό που προτείνουν αυτοί που μας κυβερνούν. Όπως έλεγε η μητέρα μου, μάρτυρας και ιδρύτρια του κινήματος η Λάουρα Πογιάν. Είμαστε μία και πολλές. Είμαστε ειρηνική φωνή, ειρηνική δράση για σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, για τη νίκη της δικαιοσύνης. Θα μας χτύπησαν μας προσέβαλαν, μας, μας έδιραν ορισμένες φορές. Αλλά η ανθεκτικότητά μας είναι μεγαλύτερη από το μίσος. Δεν θέλουμε να στηριχθούμε στην έννοια της, ε, ε, του θύματος. Στηριζόμαστε σε αυτά που είπε ο Γκάντι, ότι η, η ειρήνη είναι νίκη, είναι δύναμη. Χρησιμοποίησαμε το λευκό χρώμα, σύμβουλο αγνότητας, ειρήνης και δικαιοσύνης. Η μάχη μας είναι μη βιαιή, εξού και η πεποίθησή μας για τη νίκη. Μένει Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα για να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι απλώς μια κούβα που θα κυβερνιέται από τις ίδιες αρχές δημοκρατίας και ανεκτικότητας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για, γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας εδώ σήμερα σε αυτό το χώρο. Φέρνουμε σήμερα εδώ την φωνή των ανδρών και γυναικών όλων των πολιτικών θέσεων, φυλών της χώρας μας που συνεχίζουν να είναι στη φυλακή ή να καταπιέζονται με βίαιο τρόπο διότι σκέφτονται και δρούν διαφορετικά από την κυβέρνηση. Γιατί είμαστε το αναπόσπαστο τμήμα του λαού αυτού. Ευχαριστούμε ιδίως την αλληλεγγύη σας και την δέσμευση να πετύχουμε οι θυσίες αυτές να μην γίνουν εις Ζούμε σε μια πολύ ειδική εποχή στην ιστορία μας. Η ελεγγύη της Ευρώπης με τα βέλτιστα συμφέροντα του λαού της Κούβας είναι κρίσιμο για μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, στηριζόμαστε σε εσά. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Η Κούβα θα είναι ελεύθερη και δημοκρατική. Λάουρα Πογιάν, αφιερώνουμε σε εσένα το βραβείο αυτό, Ελευθερία για το λαό της Κούβας. Σα ευχαριστώ όλους. Ο πρόεδρο κύριο Μπροκ. Σα ευχαριστώ για τα λόγια που είπατε που μας βρίσκουν ε, όλους σύμφωνους και υποστηρικτές σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ζουλίκ, τη Επιτροπής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Κυρία Μπέρτα Σόλες, κυρία Μπέρκε Καστίγιο Ραμίδε, σα ευχαριστώ. Κόρη τη κυρία Λαμπράδα Πογιάν και την Μπιάνκα Ρέγε ε, Καστανιών και την Ελένκα Ρέγκα που τη συνοδεύουν. Τις ευχαριστώ όλε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ω Προέδρο τη Επιτροπή ανάπτυξη να λάβω το λόγο μετά από αυτή την συγκινητική ομιλία σας. Πιστεύω ότι η επιλογή που έκαναν οι συνάδελφοί μου το 2005 να απονείμουν το βραβείο Ζαχάροφ στις ε, γυναίκες με τα λευκά ήταν πολύ καλή επιλογή. Ενσαρκώνεται με λαμπρό τρόπο την ελευθερία του πνεύματος, την ελευθερία της σκέψης. Η ειρηνική σας δράση Κυρια... κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή και οι θετικές σας δράσεις στον πληθυσμό της Κούβας είναι δείγμα μέλλοντος, ειρήνης και μια μη βίαιη διαμαρτυρία κατά της πίεσης και της καταπίεσης που βιώνει εδώ και κοντά 60 χρόνια ο... Ε, εδώ και κοντά 50 χρόνια ο λαός της Κούβας χάρη σε γυναίκες και σαν και εσάς, χάρη σε άνδρες όπως οι αγαπημένοι, οι σύζυγοί σας, τα παιδιά σας, οι σύντροφοί σας, μπορούμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον της Κούβας ξέρουμε ότι το καθεστώς φτάνει στο τέλος του και η δημοκρατία και η ελευθερία είναι μπροστά σας. Ευχαριστώ για ό,τι κάνετε, ευχαριστώ για ό,τι κάνετε για όλο τον κόσμο με αυτή την ειρηνική αντίστασή σας και μπράβο για το βραβείο και ευχαριστούμε που ήρθατε μετά από τόσο πολύ καιρό. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίπ, έχετε το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια συγκινητική περίσταση αυτή, γιατί βλέποντας τις κυρίες στα λευκά να λαμβάνουν το βραβείο τους μετά από 8 χρόνια. Ένα βραβείο το οποίο τόσο πολύ αξίζουν και τόσο πολύ το επισημούσαν να το λάβουν τα, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλά μέλη από την Ισπανία, από την ε, πρώην Ανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, μέλη από την Πολωνία επίσης ε, που πιστεύουν ότι αξίζεται αυτή την ε, ε τιμητική διάκριση. Εκ μέρους λοιπόν της Υποεπιτροπής Ασπίνων Δικαιωμάτων, Επιτροπής Ασπίνων Δικαιωμάτων, σας ευχαριστώ για όλη αυτή την ενεργητικότητα, την προσπάθειά σας και με τη βοήθεια του λευκού χρώματος καταφέρατε να συντρίψετε το καθεστώς. Διασώσατε την αξιοπρέπεια των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Συγχαρητήρια και πάλι για όλα αυτά τα οποία κάνετε για το λαό της Κούβας. Ακόμα και σε στιγμές ευτυχίας όπως η σημερινή πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν ακόμα βραβευμένοι με το βραβείο Ζαχάροφ που δεν έχουν μπορέσει να λάβουν ε, το βραβείο αυτό, ε, να, το, να το παραλάβουν προσωπικά. Ο Γκουγέρμο Φαρινάς παραδείγματος χάρη, ένας από του τρεις κουβανού αποδέκτε του βραβείου. Επίσης, Ράζαν Ζαΐντα από τη Συρία το 2011. Δέκα χρόνια μετά μπορέσαμε τελικά να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα μετά από το ξέφρασμα της μαύρης άνοιξης της Κούβας. Όμως δεν έχουμε ακόμα τελειώσει. Πολλά ακόμα πράγματα ε, βασανίζουν τον κουβανικό λαό. Πιστεύουμε ο Γκουλιέλμο Φαρίνας ε, και η αποδέκτης ε, του βραβείου από τη Συρία θα μπορέσουν σύντομα να έρθουν και να παραλάβουν προσωπικά το, τη διάκριση αυτή την οποία να αξίζουν. Και εμείς ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους καλωσορίσουμε θερμά, όποτε μπορέσουν. Ευχαριστώ. Nun kommt, äh, Madame for... Η κυρία Μπόσκουατ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αγαπητές κυρίες τα Λευκά, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είσαστε μετά από 8 μακριά χρόνια και εκ μέρους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής ε, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσετε επιτέλους να επισκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πάρετε το βραβείο αυτό που σας απονεμήθηκε το 2005. Έχετε πολεμήσει για τη δημοκρατία την, τα, και τα ανθρώπινη δικαιώματα στην Κούβα. Ε, ένας αγώνας που έχει εμπνεύσει όλους. Ε, επί χρόνια κάθε Κυριακή περπατούσατε στους δρόμους της Σαββάνας για την, ζητώνε να απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Σήμερα είσαστε εδώ και εμείς ε, είμαστε μαζί σας. Η Κούβα μπορεί γεωγραφικά να είναι νησί, όμως όσον αφορά τις εξελίξεις της διεθνής δεν είναι νησί. Χαιρετίζουμε ορισμένα θετικά βήματα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνησή σας πρόσφατα όπως ε, τις ε, βίζες, θεωρήσεις που επιτρέπουν να ταξιδεύουν κουβανοί πολίτες αλλά λαμβάνονται τώρα και άλλα μέτρα μέσω του διμερούς διαλόγου και διμερών συμφωνιών με την Κούβα. Ελπίζω αυτά τα θετικά βήματα θα τα ακολουθήσουν πολλά άλλα θετικά βήματα και θα οδηγήσουν στην, στον πλήρη εκδημοκρατισμό της Κούβας. Αγαπητές κυρίες στα Λευκά, μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη υποστήριξή μας και ιδίως από την Επιτροπή μου και εμένα προσωπικά ως Πρόεδρου. Ο πρόεδρος Μπρόκ, σα ευχαριστώ πολύ και τώρα οι συντονιστές για δύο λεπτά και πρώτος ο κύριος Σαλαφράνκα για το Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως θύμισε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, το 2003 υπήρξε ένα μαζικό κύμα συλλήψεων, θύματα των οποίων ήταν οι περασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι ειρηνικοί ε, αντιφρονούντες και ανεξάρτητη δημοσιογράφοι όπως ο Ραούλ Ριβέρο που καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλακή ο φωτογράφος ο Μάρο Ροντρίγκε ή ο Ρολάντο Αρόγιο που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια. 7 χρόνια. Εμείς βάσει αυτών των ιδεών προτείναμε την βράβευση των Ντάμα Στεμπλάνκο γιατί είναι δείγμα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των λαών και μιας προσπάθειας να δώσουν φωνή στους λαούς. Στη ζωή, πρόεδρε, δεν υπάρχουν Άτομα υπάρχουν που γίνονται μάρτυρες. Δεν υπάρχουν παραδείγματα. Άνθρωποι υπάρχουν που γίνονται παραδείγματα. Τις βλέπουμε εδώ. Άτομα που καταπιέστηκαν, ε, υβρίστηκαν και που αντέχουν, προστατεύουν την, την αξιοπρέπειά τους και αγωνίζονται για την ελευθερία τη δική τους και των αγαπημένων τους. Μετά από τόσα χρόνια το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει αυτά τα γενναία άτομα που υποστήριξαν την ελευθερία και την ε, ε, αξιοπρέπεια και με συγκίνηση ακούσαμε τα λόγια που αναφέρθηκαν στη μνήμη της Λάουρα Πογιάν. Θα θυμίσω, Πρόεδρε, κάποια λόγια. Τον Οσβάλντο Παγιά ανέφερε ο Πρόεδρος. Να σας θυμίσω εγώ κάτι που έλεγε ο Οσβάλντο Παγιά στο, στο, στην Ολομέλεια. Δεν έχω μίσο στην καρδιά, αλλά αυτή που με καταπιέζουν δεν θα κυριαρχήσουν στην καρδιά μου. Είναι λόγια που είπε ο του Κοινοβουλίου και ο αγώνας αυτός είναι δικός μας αγώνας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, με μεγάλη χαρά σας ε, δέχομαι εδώ για να σας δώσουμε αυτό το βραβείο που σας δίνουμε με μεγάλη τιμή. Είστε αγωνίστρες για την ελευθερία, για τα δικαιώματα του λαού σας. Η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες, ήταν μία από τις ομάδες που στο κοινοβούλιο αυτό μόνιμα αντιτάθηκε στο εμπάργο που έχει επιβληθεί στην Κούβα γιατί θεωρούμε ότι τούτο χρησιμοποιείται ως όπλο κατά του λαού της Κούβας από πλευράς του καθεστώτος της Κούβας και δεν εξυπηρετούσε την υπόθεση της ελευθερίας. Ευτυχώς η τωρινή κυβέρνηση της Αμερικής το κατάλαβε και το ελάφρυνε. Αυτό παρεπιτρέπει να προχωρήσουν όλες οι αλλαγές που πηγαίνουν προς την υποστήριξη της μάχης εκείνων που όπως εσείς οι οικογένειές σας αγωνίζονται για την ελευθερία μόνιμα και συνεχώς με την δύναμη της πεποίθησής σας. Είμαι μία από τις πολλές και τους πολλούς στο Κοινοβούλιο που βιώσαμε δικτατορία και αξιολογούμε σημαντικά τον αγώνα για την ελευθερία. Και γι' αυτό σας λέω ότι εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, είμαστε μαζί σας. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τελειώσει η δικτατορία, για να μπορέσουν όλοι οι Κουβανέζοι να βιώσουν όλες τις ατομικές ελευθερίες. Ξέρουμε ότι οι Κουβανοί είναι έτοιμοι για την ελευθερία, είναι έτοιμοι για τη δημοκρατία όπως όλοι οι λαοί του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ για τον αγώνα σας. Θα την παρακολουθήσουμε μαζί μας και ελπίζουμε ότι θα γιορτάσουμε την ελεύθερη Κούβα. Εσείς κυρία Νέιτς, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Εδώ είμαι κυρίες με τα λευκά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων Δημοκρατών Καλώ ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από τόσα χρόνια, μετά από την απονομή του, του βραβείου Ζαχάροφ. Επιτέλους ήρθε η σημερινή μέρα ώστε να μπορέσετε να προσέλθετε εδώ για να παραλάβετε το βραβείο. Σήμερα αποτείουμε φόρο τιμής στις διαμαρτυρίες στις οποίες προέβητε υπό δυσχερείς συνθήκες, διαμαρτυρίες οι οποίες έστρεψαν τα όματα τη διεθνούς κοινή στη βαριά μοίρα των αντιφρονούντων οι οποίοι τόλμησαν να επικρίνουν την έλλειψη πολιτικών ελευθεριών στην Κούβα. Και σήμερα βέβαια τιμούμε και την μνήμη και το θάρρος της Λάουρα Ινές Πογιάν Τολέδο, της ε, θαραλέας ιδρύτριας των ε, κυριών λευκά η οποία έχει αποβιώσει. Ευτυχώς η πολιτική κρατούμενη των οποίων ε, καταδείξατε την ε, βαριά μοίρα έχουν απολυθεί. Από το 2005 ωστόσο, σε ό,τι αφορά πολιτικές ελευθερίες και δικαιώματα, δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα ή δεν έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχει βελτιωθεί μεν ελαφρά, αλλά όχι επαρκώς. Και για το λόγο αυτό οι διαμαρτυρίες σας συνεχίζονται. Και κάθε μέρα περισσότερες γυναίκες προσέρχονται και πυκνώνουν τις γραμμές των κυριών με τα λευκά που δείχνει ότι το μήνυμά σας ειρήνης και διαμαρτυρίας εξακολουθεί να είναι το ίδιο σημαντικό και επίκαιρο όπως ήταν το 2005. Σύμφωνα με το Human Rights Watch η Κούβα είναι από τις λίγες χώρες στην ε, ή και η μόνη χώρα στη Λατινική Αμερική η οποία παρεμποδίζει κάθε ε, μορφή πολιτικής πρόοδου και είναι πραγματικά κρίμα που από τους πολιτικούς κρατουμένους οι οποίοι συνελήφθησαν επί Φιντελ Κάστρο παραμένουν στις φυλακές. Ο δε νυν πρόεδρος Ραούλ Κάστρο χρησιμοποιεί ε, τους ε, καταπιστικούς νόμους που δίνουν το δικαίωμα να κάνει συνοπτικές δίκες για να καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο το μόνο φωτάκι στο τέλος του τούνελ είναι ότι ο πρόεδρος ήρε εν μέρη την πεντα, από πεντηκονταετία στις απαγόρευση εξόδου από τη χώρα των ίδιων κουβανών πολιτών. Κάτι που επέτρεψε και σε εσά βεβαίω να έρθετε εδώ να παραλάβετε το βραβείο που δικαίως σας απονεμήθηκε και για το οποίο σας συγχαίρουμε εκ, εκβάθους ε, εκ βάθους καρδίας. Τάνοκ, ομάδα ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Ντάμαστε Μπλάνκα, εδώ βρίσκομαι. Και εγώ λοιπόν εξ ονόματος της ομάδας μου των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών σας συγχαίρω. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μετά από 8 χρόνια, γιατί εγώ τότε προείδρευα της Ολομέλειας όταν έγινε η απονομή του βραβείου, ήρθατε λοιπόν και μπορέσατε να παραλάβετε το βραβείο του 2005 έτσι λοιπόν έφτασε στα χέρια των ε, προσώπων που πραγματικά ε, το αξίζουν. Η Κούβα εξακολουθεί να είναι μια βάρβαρη κομμουνιστική δικτατορία για μας. Παρά τις υποσχέσεις που έχει κάνει ο Ραούλ Κάστρο και βέβαια κάποιες περιορισμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις έγιναν, ωστόσο δεν ακολουθούνται από πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ούτε από τον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι η Κούβα παραμένει η μόνη χώρα στη Λατινική Αμερική η οποία παρεμποδίζει οποιαδήποτε κριτική κατά του καθεστώς, σύμφωνα με την Human Rights Watch, και παραμένει από τις πιο καταπιστικές χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι ε, δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα στην έκθεσή τους λένε ότι από 179 χώρες του πλανήτη η Κούβα είναι στην 171η θέση σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου. Ακόμα δεκάδες ή εκατοντάδες κρατούμενοι αναμένουν δίκη. 126 πολιτικοί κρατούμενοι απολύθηκαν τα έτη 2010 και 2011, αλλά μετά από πίεση και μεσολάβηση της Καθολικής Εκκλησίας και της Ισπανικής Κυβερνήσεως. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν, χωρίς να αρθούν οι κατηγορίες. Περιέργως, η ε, Κούβα εξακολουθεί να είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εξ ονόματος της ομάδας μου λοιπόν, αλλά είμαι και στην Υποεπιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, απευθύνω χαιρετισμό στο θάρρος και στον αγώνα σας από τις, ε, τις ε, κυρίες στα Λευκά. Με, λίγα, με τα λίγα ισπανικά μου θα πω Ζήτω η ελεύθερη δημοκρατική Κούβα. Δεν μπορεί να κυβερνά ο Κάστρο για πάντα. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες με τα λευκά. Χαίρει και η δική μου πολιτική ομάδα για το γεγονός ότι οι κυρίες με τα λευκά μπόρεσαν να έρθουν από την Κουβά εδώ για να παραλάβουν το βραβείο τους. Εσείς αγωνίζεστε για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Όμως στην Κούβα και κάτω από διαφορετικές συνθήκες από ό,τι αγωνιζόμαστε εμείς εδώ. Εμείς νομίζω δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ποιες είναι οι συνθήκες στην χώρα σας. Σας υποστηρίζουμε λοιπόν με το βραβείο Ζαχάροφ στην προσπάθειά σας και απευθύνω και τις προσωπικές μου ευχές για τον αγώνα σας αυτό. Έχει έρθει η ώρα να γίνει η, να έρθει η ελευθερία στην Κούβα. Διότι γνωρίζω ότι εκεί εξακολουθούν, εξακολουθεί να ισχύει καταπιστικό καθεστώς, οι δε μεταρρυθμίσεις προχωρούν βραδύτατα εντυπωσιάστηκα από την την ε, περιγραφή του blogger Sanchez στην Κούβα που λέει ότι με παρακολουθούν διαρκώς. Πρόκειται για απολυταρχικό καθεστώς που μπορεί να καταστρέψει την κάθε πτυχή της ζωής του κάθε ατόμου από την οικογενειακή με την επαγγελματική. Αυτή είναι η παράθεση που ήθελα να κάνω. Αγαπητές κυρίες με τα λευκά, όσο διατηρείται το καταπιστικό καθεστώς στην Κούβα, εμείς από την Ευρώπη θα υποστηρίζουμε το, την άλλη Κούβα που για μας έχει υπαρξιακή σημασία. Η κυρία Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, σήμερα είμαστε εδώ οι κυρίες με τα λευκά. Όχι επειδή έδειξε καλή βούληση, καλή προαίρεση η κυβέρνηση της Κούβας, αλλά ε, διότι υπήρξαν πολιτικές πιέσεις, διότι είμαστε, είναι αποτέλεσμα της ελπίδας τόσων ετών. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δεχθούμε το βραβείο Ζαχάροφ βραβείο που άντρες και γυναίκες στο κοινοβούλιο εμπιστεύτηκαν σε μας. Πρέπει να ξέρετε κύριε Πρόεδρε ότι οι κυρίες με τα λευκά δεν θα προόδωσουμε, δεν θα σας εξαπατήσουμε. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Ο αγώνας μας είναι ένας ειλικρινής αγώνας. Ένας αγώνας που κάνουμε με ειρηνικό τρόπο, διότι είμαστε γυναίκες που αγαπούμε την οικογένεια. Είμαστε γυναίκες που αγαπούμε τη ζωή. Είμαστε όμως γυναίκες που μάθαμε πολλά για την ε, χώρα μας και ο αγώνας συνεχίζεται. Ευχαριστούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δεν μέχρι ότου έχουμε ελεύθερους τους δικούς μας, αλλά και κυρίως όταν έχουμε μία νέα κούβα που υπάρχει δικαίωμα ανθρωπίνο, ανθρώπινο δικαίωμα, όπου μια κούβα χωρίς τους κάστρο κύριος. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Μπροκ, αγαπητές κυρίες με τα λευκά, σας συγχαίρω και πάλι για το βραβείο και να σας ευχαριστήσω για τα όσα έχετε πράξει και υπό την ηγεσία της Λάουρα Πολάν από την Μαύρη Κοινή Άνοιξη του 2003 έχετε αποδείξει μέγα θάρρος. Βρήκαμε τα ίδια λόγια, εσείς και εμείς, ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Για μας δεν κοστίζει τίποτα να μην πούμε τα λόγια αυτά. Για εσά ναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και αυτό σημαίνει ότι δείξατε μέγιστο θάρρος που εμείς δεν θα χρειαστεί νομίζω να αποδείξουμε ποτέ. Αυτό σας κάνει τόσο μοναδικές στο έργο σας και γι' αυτό γίνεστε και σύμβολο για μας. Γιατί καμιά φορά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν στρέφονται όλα γύρω από τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πρέπει να δούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να παίζουν κέριο ρόλο. Είπαμε ότι η κουβανική ηγεσία ξεκίνησε κάποιε οικονομικέ μεταρρυθμίσει και λόγω τη δυσχερέστας τη οικονομική καταστάσεω. Γνωρίζουμε από την ευρωπαϊκή μα ιστορία, ωστόσο, ότι η πραγματική κοινωνική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη για του ανθρώπου μπορεί να υπαρξει μονο μόνον εφόσον βαδίζει χέρι-χέρι με την δημοκρατία και την ελευθερία. Πρέπει λοιπόν να πληρούνται οι συνθήκε αυτέ και μόνο τότε ε, μπορεί να είναι εξασφαλισμένο αυτό. Τα νούμερα που δεν γνώριζα και τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος Σούλτς με κατέπληξαν. Δεν τα γνώριζα. Διαπιστώνω ότι στα θέματα ελευθερίας δεν έχουν επιτευχθεί πραγματικά βήματα πρόοδου. Δύο φορές η χώρα μου πέρασε από απολυταρχικά καθεστώτα. Είναι πάντοτε κρίσιμο να μην υπάρχει μονάχα ένα κόμμα η θράψη αυτού του μονοκαματικού καθεστώτος έχει κέρια σημασία. Να μπορούν να επιλέξουν οι άνθρωποι, να μπορούν να ανταγωνίζονται οι πολιτικοί για να προσελκύσουν τους, τις ψήφους των ανθρώπων. Αυτό μέσα στα πλαίσια μιας γενικής προσπάθειας σε όλη την Ελληνική Αμερική. Να ξεπεραστούν επιτέλους. Είτε οι δεξιές είτε οι αριστερές δικτατορίες. Καμία διαφορά δεν έχουν. Ελπίζω στη βάση αυτή να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για, μας, για μένα σήμερα είναι ωραία, είναι όμορφη μέρα. Ήδη το 2005 ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και παρά τις πλείονες προσκλήσεις που είχα από την Κούβα δεν πήγα ακριβώς διότι δεν είχε απονεμηθεί και παραληφθεί, δεν είχε παραληφθεί από εσά το βραβείο. Σήμερα είμαι πια ελεύθερος να μεταβώ στην Κούβα.